Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε για να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας με 10 λεπτά καθυστέρηση και ζητώ συγγνώμη από τους διερμηνείς κυρίως, λέει ο Μιλήτρια, η Πρόεδρος. Έχετε την ημερήσια διάταξη, δεν ε, έχει ζητηθεί καμία τροποποίηση, συνεπώς εγκρίνεται. Ανακοινώσεις. Τέσσερις έχω. Πρώτον, υπάρχει διάσκεψη για την απασχόληση των νέων, που έγινε τελικά κάτι σαν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έλαβε χώρα στο Παρίσι προχτές και εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρό μας, τον Μάρτιν Σούλτς. Ο Μάρτιν Σούλτς Μάλιστα μου ζήτησε να το συνοδεύσω. Οπότε και εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών ε, Υποθέσεων πήγα και εγώ μαζί του για να εκπροσωπήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκεί. Είχαμε πρώτα λοιπόν στο Παρίσι πρώτα μια συνάντηση των Υπουργών Απασχόλησης και Εργασίας και κατά αυτή τη συνεδρίαση πήρα και εγώ το λόγο. Ανέφερα πώς προχωρούν οι δικές μας εργασίες και ανέφερε και τις ανησυχίες που εκφράζονται εδώ, σε αυτήν εδώ την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κυρίως μάλιστα το γεγονός της ανεργίας των νέων που δεν μπορεί να λυθεί μόνο με την κινητοποίηση. Η κινητοποίηση πρέπει να οργανωθεί σε θελοντική βάση, καταρχήν. Υπενθύμησα επίσης από την εμπειρία και από το μέχρι τώρα έργο μας γνωρίζουμε ότι η εγγύηση για τους νέους, το πρόγραμμα αυτό δηλαδή και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων δεν θα πετύχουν παρά μόνο εάν στηρίζονται στις βέλτιστες πρακτικές όπως λέγονται. Δηλαδή να υπάρχει άμεση συνεργασία των κοινωνικών εταίρων κάθε φορά που τίθενται σε εφαρμογή τέτοιου είδου προγράμματα. Υπογράμμισα επίσης την σημασία που δίνουμε, πέρα από την πρωτοβουλία αυτή δηλαδή για την απασχόληση των νέων, στα στοιχεία τα οποία επιτρέπουν ανάκαμψη της οικονομίας και στις χώρες της περιφέρειας, όπως επίσης και τη σημασία που δίνουμε στην εταιρική σχέση προκειμένου να πάρουν στα χέρια τους το μέλλον τους οι νέοι. Ότι θέλουμε και αυτά να στηριχθούν εξίσου ναι η Τραπεζική Ένωση, αλλά ναι και σε οτιδήποτε ενισχύει την, ε, τις νέες οι μικροπιστώσεις, η κατάρτιση κλπ. Ανέφερα και δύο ακόμα σημεία. Πρώτον, υπογράμμισα ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας κάθε φορά που ασχολούμαστε με την απασχόληση των νέων, το ότι υπάρχουν διαφορές πολύ μεγαλύτερες μάλιστα ίσως ε, σήμερα μέσα στην Ευρωζώνη σε σχέση με έξω από την Ευρωζώνη και ζήτησα από τους υπουργούς εφεξής να κινητοποιηθούν όλοι προκειμένου να δώσουν το δικό τους ο καθένας πρόγραμμα εργασίας. Γιατί όπως ξέρετε, προκειμένου τα προγράμματα αυτά να είναι αποτελεσματικά, πρέπει να υιοθετήσουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, να υιοθετήσουμε την, τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα κράτη-μέλη από τη δικιά τους την πλευρά να δώσουν το δικό τους πρόγραμμα εργασίας. Ενώ από όσο ξέρω, τι από όσο ξέρω, είναι γεγονός, μόνο έξι χώρες έχουν δώσει τα δικά τους εθνικά προγράμματα μέχρι σήμερα. Και οι έξι αυτές χώρες είναι η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Λετωνία, η Πολωνία και η Σλοβακία. Τους είπα λοιπόν ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν τα προγράμματα αυτά, ε, οι χώρες μέλη να τα δώσουν, να μας τα στείλουν. Επίμενα, επέμεινα βέβαια πολύ σε αυτό, γιατί όταν πήγαμε στην Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα, συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Απασχόλησης εκεί και με ξέπληξε. Τον ρώτησα πού βρίσκεστε όσον αφορά το δικό σας πρόγραμμα εργασίας για την εγγύηση των νέων και για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Τι μου απάντησε, μου είπε, ε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη διάσκεψη των Παρισίων. Ε, νομίζω ότι εδώ στρεβλώνονται τα πράγματα, τι έρχεται πρώτο δηλαδή και τι δεύτερο. Τώρα για τη διάσκεψη αυτή υπήρχαν 24 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πήρε το λόγο και είπε πόσο μεγάλη σημασία έχει η προτεραιότητα αυτή για τους νέους, δίνοντας την εξή εικόνα, είπε οι γονεί μα, οι δικοί μα οι γονεί, ήταν μια γενιά που αναγκάστηκε να κάνει πάρα πολλέ προσπάθειες. Οι προσπάθειε όμω που έπρεπε να κάνουν ήταν στο όνομα του μέλλοντος. Κινητοποίηση για την ανοικοδόμηση των διαφόρων χωρών για τα παιδιά τους. Ενώ τώρα σε αυτήν τη γενιά τι ζητάμε από αυτούς. Ζητάμε να σωθούν οι τράπεζες. Είπε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο δεν περνάει καλά. Αν λοιπόν ε, πούμε ανταυτού στους γονείς ότι πρέπει να κοινοτοποιηθούν για να σώσουν το μέλλον των παιδιών τους, ίσως τότε να ε, περάσει πιο εύκολα το μήνυμά μας. Πολλοί τον ρώτησαν πότε θα ψηφίσει τέλος πάντων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ο πρόεδρος Σούλς είπε ότι τα χρήματα θα αποδεσμευθούν 20 Νοεμβρίου καταρχήν, δηλαδή μετά την Ολομέλεια του Στρασβούρου. Οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων επίσης πήραν το λόγο. Και ανάμεσα στις πιο δυνατές παρεμβάσεις, σημειώνω εγώ εκείνη του Ιταλού ε, Προέδρου, του Ενρίκο Λέτα, της Ιταλικής Κυβέρνησης, ο οποίος αναφέρθηκε στην επόμενη διάσκεψη που θα γίνει τον Απρίλιο Τώρα εκεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξε ένα ζήτημα, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει αρχές Απριλίου να γίνει μια διάσκεψη για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη θα θέσουν σε εφαρμογή την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και ο πρόεδρος Λέτα θα οργανώσει πάλι τον Απρίλιο λίγο αργότερα στη Ρώμη για να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα πριν από τις ευρωεκλογέ για να κινητοποιήσει τον κόσμο πάλι με αυτή την ιδέα. Το Βερολίνο αποφασίσαμε την αρχή, στο Παρίσι τα μέσα και στη Ρώμη θα γίνει ένας πρώτος γύρος τραπεζιού για να δούμε τελικά τι έχουμε αποφασίσει και πώς προχωράμε. Επίσης, ο Φιλανδός ηγέτης αναφέρθηκε στους μηχανισμούς που έχουν εκείνη θέση σε εφαρμογή και ενημέρωσε έτσι τις άλλες χώρες μέλη. Ένα άλλο θέμα το οποίο τέθηκε είχε να κάνει με την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Εκεί είχαμε παρέμβαση του Έλιο Ντιρούπου, του Βέλγου Πρωθυπουργού, ο οποίος υπογράμμισε ότι πέρα από το θέμα της ανεργίας των νέων υπάρχει και το θέμα του dumping, δηλαδή των συνθήκων εργασίας, της ποιότητας της απασχόλησης που προσφέρεται στους νέους, ότι και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε, ολοκληρώνοντα την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Και ρώτησε από αυτό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει πού βρισκόμαστε. Ο πρόεδρο Παρόσο, που βρισκομαστε ο προεδρος παροσο που κληθηκε να απαντήσει, είπε ότι το μπαλάκι είναι στο Συμβούλιο. Ότι το Συμβούλιο πρέπει να συμφωνήσει στο επόμενο Συμβούλιο Εύσκο Κοινωνικών Υποθέσεων. Και ο πρόεδρος Φανραπόη ολοκλήρωσε τις εργασίες λέγοντας ότι αν το Συμβούλιο αυτό δεν καταφέρει να πετύχει συμφωνία, τότε το θέμα αυτό θα εξεταστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πια. Και για να ολοκληρώσω, έχω να προσθέσω τα εξή δύο. Πρώτον, πολλοί συζήτησαν για το θέμα μιας ε, κοινοτικής αρμοδιότητας ουσιαστικά που συζητιέται σε επίπεδο χωρών μελών. Δηλαδή, εφόσον είναι κοινοτικό το θέμα, γιατί το συζητάει ένα σχήμα το οποίο θυμίζει περισσότερο Συμβούλιο Υπουργών. Όμως πρέπει να υπάρχει μια καλή δυναμική όταν εξετάζεται το θέμα αυτό και από πλευρά των χωρών μελών, γιατί την αρμοδιότητα την έχουν πρώτα τα κράτη-μέλη. Οπότε, ναι μεν υπήρξε εκεί ένα ζήτημα, αλλά ο πρόεδρος Φαν Ρομπά συμφώνησε απόλυτα με το όλο εγχείρημα. Και ο πρόεδρος Ολάντ κατέληξε στα συμπεράσματα λέγοντας ότι τώρα πρέπει όλοι να δώσουν το πρόγραμμα εργασία τους, όλες οι χώρες δηλαδή, ότι πρέπει να έχουμε ένα ποιοτικό πλαίσιο προκειμένου να οργανωθεί αυτή η ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και ότι οι προτάσεις οι οποίες έγιναν και θα γίνει και στη συνέχεια πρέπει να είναι ποιότητας. Αυτά είχα να σας πω σε σχέση με τη διάσκεψη αυτή που έλαβε χώρα στο Παρίσι. Η δεύτερη μου ανακοίνωση είχε να κάνει με κάτι άλλο. Στην επόμενη συνεδρίασή μας, δηλαδή 25 και 26 Νοεμβρίου, 26 Νοεμβρίου το απόγευμα δεν θα συνεδριάσουμε. Ακυρώθηκε ή θα ακυρωθεί τέλο πάντων. Άρα είσαστε ελεύθεροι το απόγευμα. Τρίτη παρατήρηση. Όσον αφορά την ε, Γερμανία που δεν χρησιμοποιείται, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα η επιθεώρηση αυτή που γίνεται βελτιώνει τα πράγματα. Σας ευχαριστώ. Τέλος, σύμφωνα με την συνήθη πρακτική μας, σας υπενθυμίζω ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται μέσω διαδικτύου. Μπορεί κανείς να την παρακολουθεί στο διαδικτύο. Και τρίτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, πρακτικά 18 Σεπτεμβρίου τα έχετε. Αν δεν έχουμε σχόλια, θεωρούνται εγκεκριμένα. Est-ce que Έρχομαι τώρα στο σημείο 4. Ο κύριος Νταρντέν έχει πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε το σημείο του μετά τις ψηφοφορίες για να μπορέσουμε να τηρήσουμε την ημερήσια διάταξη, το χρονοδιάγραμμα της ημερήσιας διάταξης, θαυμάσια. Σημείο 6 λοιπόν και δίνω το λόγο στον Αλεχάνδρο Θέρκας για να μας πει ποια είναι η κατάσταση των συζητήσεων και το αποτέλεσμα των ανταλλαγών απόψεων σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο για τις ε, συνθήκες ε, εισόδου και διαμονής και εγκατάστασης των ε, υπηκών τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχει υπερατωθεί πια αυτή η επεξεργασία ενός από τα σημαντικότερα θέματα σε αυτή τη θητεία. Ο κύριος Κομφεράτη θα πρέπει να παρουσιάσει τα θέματα επί της ουσίας. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να μπορέσουμε να κλείσουμε τη διαδικασία αυτή μετά από τον κύριο Μαρτίνες ε, για αυτό το θέμα που απασχόλησε το Συμβουλίο, την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο σε πάρα πολλούς τριγωνικούς διαλόγους. Ο τελευταίος έγινε στις 23 Οκτωβρίου και καταλήξαμε σε συνολική συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου με την θετική γνώμη και της Κομισιόν. Αυτή η συμφωνία επίσης επικυρώθηκε από την Κορεπέρ. Διακόπτη η πρόεδρος. Χωρίς μικρόφωνο η πρόεδρος. Τι να κάνω. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. επαναλαμβάνω. Βρισκόμαστε στο τέλος μιας μακράς πορείας και μιας μακράς εργασίας στην Επιτροπή μας που στέφεται υπό επιτυχία πια και θα ήθελα να σας πω ότι ο αρμόδιος για όλα αυτά που αξίζει την ε, του επένου μα ήταν ο Σέρχιο, Σέργιο Κομφεράτη που εργάστηκε για πάρα πολύ καιρό για το θέμα αυτό και η κυρία Μαρτίνες και εγώ επίσης βοηθήσαμε στο τελευταίο τμήμα της εργασίας αυτής στον ε, τριγωνικό διάλογο που έγινε στις 23 Οκτωβρίου που κατέληξε και σε μια συνολική συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Είχαμε και μια συνάντηση προηγουμένως με τους κοιόδης εισηγητές οι οποίοι και αυτοί συμφώνησαν με την θέση του Συμβουλίου. Η συμφωνία αυτή επίση ενεκρίθη από την συνεδρία της Κορεπέρ τη ΜΕΑ στα τέλη Οκτωβρίου και έτσι έχει τελειώσει η διαδικασία <clears throat> και παραμένει μονάχα το θέμα τη κοινοβουλευτική ε, ψηφοφορία για να εγκριθεί αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε αυτά τα απορίσματα των διαπραγματεύσεων γιατί έχουμε επιτύχει όλου του στόχου που είχε η Επιτροπή Απασχόληση. Είχαμε <clears throat> αποκλειστική αρμοδιότητα για το άρθρο 50 και σε άλλα δύο άρθρα όπως είναι το 17 και διάφορες αιτιολογικές σκέψεις. Όλα αυτά μέσα στα πλαίσια μιας ε, κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ ημών και της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπήρχε η ίδια, μεταχείριση στα εργασιακά θέματα και σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας ώστε οι εποχιακοί εργαζόμενοι να μην έρχονται στις χώρες υποδοχής σε υποδέστες συνθήκες από τους εθνικούς εργαζόμενους. Αυτή ήταν η βασική φιλοσοφία της Επιτροπής μας, να εξασφαλίσουμε ότι θα υπήρχε ισότης μεταχείρισης με τους εθνικούς εργαζόμενους για να μην υπάρξουν φαινόμενα εκμετάλλευσης και να μην αναζηροποιηθεί ο ρατσισμός και η ξενοφοβία στην Ευρώπη. Αυτό το στόχο λοιπόν νομίζω τον έχουμε πετύχει απόλυτα και σε ό,τι αφορά το εργασιακό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις, όπως και σε όλες τις πτυχές κοινωνικής ασφάλειας, Απλώς θέλω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις για το Συμβούλιο. <clears throat> Έχει γίνει δεκτό να μπορούν να κάνουν εξαιρέσεις τα κράτη-μέλη για λόγους ανεργίας, προστασίας της οικογένειας και εκπαίδευσης και κατάρτισης όταν δεν είναι για επαγγελματικούς σκοπούς, αλλά είναι πάρα πολύ περιορισμένες αυτές οι εξαιρέσεις για πολύ σύντομες διαμονές στις χώρες ε, υποδοχής, ώστε για σύντομες μονάχα ε, διαμονές να μην μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία παροχής επιδομάτων ενεργείας ή οικογενειακών επιδομάτων. Και έτσι λοιπόν όλα ε, παραμένουν σε επίπεδο δυνητικό. Τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν αυτές τις εξαιρέσεις. Κατά τα άλλα υπάρχει απόλυτη ισότηση μεταχείρισης. Πιστεύω λοιπόν ότι μετά από όλα αυτά αγαπητοί συνάδελφοι έχουμε φέρει σε πέρας απόλυτα την, εντολή, την εντολή μας και χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη μπορώ να πω από τη δική μου πλευρά ότι είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και νομίζω ότι έχουμε κάνει και μια σημαντική συμβολή με την έγκριση αυτής της οδηγίας γιατί αυτή η οδηγία επιτρέπει να απελευθερωθεί και η οδηγία για τους ε, ε, εργαζόμενους που μεταφέρονται από μία επιχείρηση σε μια άλλη. Μάλλον σε, μεταξύ διαφορετικών κλάδων της ίδιας εταιρείας. Επειδή τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά για, το, για την ε, οδηγία αυτή όπου υπάρχουν πολλές δυσκολίες μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και Κοινοβουλίου τουλάχιστον αν περάσει η οδηγία για τους εποχιακούς εργαζομένους θα έχουμε τουλάχιστον ένα νομοθέτημα που θα επιτρέψει μια ισοδίκαια αντιμετώπιση αυτών των εργαζομένων που είναι χιλιάδες και χιλιάδες εργαζόμενοι οι οποίοι θα καλυφθούν από αυτήν την ρύθμιση και θα εξασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια και την ίση μεταχείρισή τους στις χώρες υποδοχής. Αυτά κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελε κάποιος να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Κυρία Εσαγιά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Κοφεράτη αλλά και τον κύριο Σέργας ε, για την πολύ καλή τους δουλειά. Ε, επικαιροποιήθηκαν οι πληροφορίες που είχαμε ε, από την τριμερή συνάντηση που έγινε με το Συμβουλίο και νομίζω όλοι, και αυτό είναι καλό, έχουμε την αίσθηση ότι οι πληροφορίε πράγματι μας δόθηκαν χωρίς καθυστέρηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Επίσης είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα γιατί όπως είπε και ο κύριος Σέρκας πλέον δεχόμαστε την ίση μεταχείριση και την κοινωνική ασφάλιση που έχουν άμεση σχέση με την προσφερόμενη εργασία. Τα θέματα της ε, κοινωνικής ασφάλισης ε, αναφέρθηκαν, τα επιδόματα για την ανεργία, τα οικογενειακά επιδόματα, τα εκπαιδευτικά συστήματα, όλα αυτά κυρίως ε, σε χώρες όπου έχουμε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που συνδέονται άμεσα με την παραμονή, νομίζω ότι αν δεν επιτυγχάναμε τη διεύνηση θα δημιουργεί το πραγματικά πρόβλημα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ικανοποιητικό και το δεχόμαστε όλοι. Επίσης, με το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε Νομίζω ότι μπορούμε πλέον να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου ένας υπήκος τρίτης χώρας θα είχε ενδεχομένως πιο ευνοϊκή θέση από υπήκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος εργαζίζεται σε άλλη χώρα από την πατρίδα του. Είναι σημαντικό να έχουμε και αυτή την αρχή κατά νου, ότι δηλαδή οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν πρέπει να έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση από τους υπηκόους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για άλλη μια φορά λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την αγαστή συνεργασία. Ε, ενδέχεται να πω και αυτό ότι σε ορισμένε χώρες ε, σήμερα η γραφειοκρατία να έχει υποχωρήσει. Αυτή είναι και η υπεραξία που επιδιώκουμε. Ίσως κάποιοι συνάδελφοί μου να το αμφισβητούν αυτό, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές, ένα σχετικό τονισμό. Και αν σε κάποιες χώρες υπάρχουν ευνοϊκότερες μεταρρυθμίσεις για τους εποχιακά εργαζόμενους, προφανώς ε, και αυτό θα είναι δυνατόν να διατηρηθούν αυτές, όπως σημαίνει πάντα και με οποτεδήποτε θεσπίζουμε διατάξεις, οδηγίες για επικόους τρίτων χωρών. Ευχαριστώ πολύ και τους άλλους και όδης εισηγητές. Κύριε Πεταμιάς, ευχαριστώ πολύ. Εν συντομία. Και εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ θετική συμφωνία, μια πολύ ε, ισορροπημένη, εξισορροπημένη συμφωνία και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ για τη συντομία σας. Κυρία Ευχαριστώ. Η δική μου θέση είναι κάπως διαφοροποιημένη στο θέμα αυτό. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια οδηγία η οποία, αντίθετα από ό,τι είπαν ορισμένοι συνάδελφοι, δεν οδηγεί σε ίση μεταχείριση των εποχιακών εργαζομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτών που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο άρθρο 12 που αναφέρεται η αποζημίωση δεν είναι σαφές τι είδους αποζημίωση θα είναι και επί τη βάση ποιων αρχών θα χορηγείται και τι είδους, τι ε, επίπεδο θα είναι αυτή η αποζημίωση. Επομένως, οι εποχιακοί εργαζόμενοι από τα νέα κράτη-μέλη είναι σε υποδέστερη θέση γιατί δεν έχουν την ίδια αποζημίωση. <clears throat> Επίσης το άρθρο 14, εδώ έχουμε μια αμφιλεγόμενη διάταξη, γιατί αυτό το οποίο προτείνεται εδώ ότι είναι ότι θα δίδεται επαρκής και υποχρεωτική στέγαση στους εργαζομένους αυτούς. Ενώ στην οδηγία για τους εσωτερικούς εποχιακούς εργαζομένους, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό πάλι είναι μια ε, ανισομέρεια σε σχέση με τη μεταχείριση των εποχιακών εργαζομένων από μέσα και από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι οι διοικητικές υποχρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται εδώ θα αποτελέσουν ένα βάρος και ένα εμπόδιο για την ε, μετακίνηση και την ομαλή ροή εποχιακών εργαζομένων από, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα δυσκολευτώ πολύ να υπερψηφίσω αυτές τις διατάξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τζιν Λάμπερτς. Κυρία Γιασλοβέξα, σας υπενθυμίζω όμως ότι το άρθρο αυτό είναι ένα άρθρο για το οποίο η Επιτροπή μας δεν είναι infine αρμόδια, διότι υπάρχει επιμερισμένη αρμοδιότητα με την ΛΥΜΠΕ. Οπότε πρέπει να τα πείτε αυτά και στον κύριο Κλοντ Μωράης που είναι συγητής της ε, Λίμπε και όχι στον κύριο Σέρκας. Ζιν Λάμπερτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με το αποτέλεσμα, αλλά θέλω να αναφερθώ λιγάκι και στο θέμα της ίσης μεταχείρισης ή όχι οι Ευρωπαίοι υπήκοοι έχουν κάποιες δυνατότητες να αλλάξουν εργοδότη, να μετακινηθούν κτλ. Κάτι το οποίο δεν δικαιούνται οι υπήκοοι τρίτων χωρών. Επανέρχομαι και σε αυτό που είπε ο Πρόεδρος, ότι τα δύο άρθρα που αναφέρθηκαν, που έχουν να κάνουν με τις κυρώσεις, τους εργοδότες και τα λοιπά που εξετάζουμε μαζί με την ΛΥΜΠΕ, θέλουμε να δούμε πώς θα ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία. Ίσως αξίζει τον κόπο να αναμίξουμε εδώ τους εθνικούς βουλευτές. Αν θέλουν να κάνουν κάτι θετικό για την ίση μεταχείριση, τότε αυτό πρέπει να ισχύει και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι ίδιες προδιαγραφές δηλαδή πρέπει να ισχύουν και διασυνοριακά. Κύριε Σιγητά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το έχω κάνει και πριν, αλλά και τώρα που άκουσα τις παρεμβάσεις των συναδέλφων, των σκιωδών εισηγητών, τους ευχαριστώ για το δικό τους έργο. Βοήθησαν πολύ και ήταν πολύ ευχάριστη η συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας. Πολύ στενή, ακούσαμε ένας τον άλλον και έτσι και για μένα η εμπειρία αυτή ήταν πολύ ευχάριστη και σας ευχαριστώ. Θέλω επίσης να διαβεβαιώσω την κυρία Γιανοβέσκα και όσους έχουν κάποια προβλήματα με άρθρα της ΛΥΜΠΕ, ναι, είμαστε εκτός αρμοδιότητας. Αυτά πρέπει να τα πείτε σε άλλες επιτροπές. Πάντως είναι μια δουλειά που έγινε από κοινού σε συμφωνία με το ΕΛΚ στη ΛΥΜΠΕ. Δηλαδή και οι δύο επιτροπές συνειδητοποίησαμε ότι έπρεπε να καταλήξουμε σε μία όσο γίνεται ευρύτερη συμφωνία, ε, συνένεση για να πάμε στο Συμβούλιο Εννοείται κανένα δεν είναι ικανοποιημένο 100% από τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, γιατί τότε δεν θα έχει νόημα. Το ΕΛΚ, η Πράσινη, η Γκουε και εμεί κάναμε κάποιε υποχωρήσει. Το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ ικανοποιητικό όμω. και εσείς ως εισηγήτρια για την απόσπαση νομίζω ότι μπορείτε να συμφωνήσετε ότι αν κάνουμε αυτό το βήμα θα ξεμπλοκάρουν τα πράγματα. Δεν έχουμε τα πάντα. Πάντως η κυρία Γιασνοβιέσκα να μην αισθάνεται το άσχημο παπάκι γιατί πρόκειται για μια συνένεση στην οποία καταλήγουμε και είναι καλή για όλους. Ευχαριστώ. Σε λίγο θα ψηφίσουμε. Οπότε ξεκινάμε τις ψηφοφορίες. Με μια μικρή καθυστέρηση και πάλι ζητώ συγγνώμη σε όσους μας παρακολουθούν. Στο σημείο 7 έχουμε την γνωμοδότηση για την Επιτροπή Προϋπολογισμών Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Είναι αίτηση από την επιχείρηση Βέστας της Δανίας. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έχετε την κάρτα σας όλοι. Πέρασε τις ψηφοφορίες. 29 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται. Δεύτερη γνωμοδότηση πάντα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Εδώ πρόκειται για αίτηση τη Νόκια από τη Φιλανδία. Ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 29 υπέρ, κανείς κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται και αυτό το κείμενο με λίγο διαφορετικό αποτέλεσμα στην ψηφοφορία. Σημείο 9. Άλλη μια περίπτωση κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση μετά από αίτηση τη επιχείρηση First Solar από τη Γερμανία. Ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. 28 υπέρ, μία ψήφος κατά, καμία αποχή. Και εγώ δεν ψήφισα. Ξέχασα, λέει πρόεδρος. Σημείο 10. Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονή υπηκών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή απασχόληση. Ο εισηγητή μα, ο Αλεχάνδρο Σέρκας, μόλις μας παρουσίασε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Ψηφίζουμε λοιπόν το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι, πέρα τη ψηφοφορίας. 26 υπέρ, μία ψήφος κατά, λέει πρόεδρο. Α, όχι, διορθώνει. 28 υπέρ, μία ψήφος κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο 11. Εδώ ψηφίζουμε το σχέδιο σύστασης. Τη συναδέρφου μας, Ίνες Σούμπερ για την εξοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη σύμβαση τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία του 2011 σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό. Σύμβαση αριθμό 189 του Διεθνού Οργάνωση Εργασία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν το σχέδιο αυτό σύσταση. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορίες. 28 υπέρ, κανείς κατά, δύο αποχές. Ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού περιεχομένου, ηλεκτρονικά και πάλι, ψηφίστε. πέρα της φοφορίας. 27 υπέρ, κανείς κατά, δύο αποχές. Συγχαρητήρια στην συντακτριά μας. Και φτάνουμε στο σημείο 12. Και εδώ πρόκειται για σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Η συνάδελφος Γιούτα Στάινρουκ είναι η συγγήτρια. Πρόκειται για τη Σύμβαση αριθμό 170 που επιτρέπει στα κρατη να κυρώσουν προς το συμφέρον της Ένωσης τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 1990 για την ασφάλεια κατά την χρησιμοποίηση των χημικών προϊόντων στην εργασία. Ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου σύστασης ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις φοφορίες. 29 υπέρ, καμία ψήφος κατά και μία αποχή. Τώρα το σχέδιο νομοθετικού περιεχομένου. Ψηφίστε. Πέρα της ψηφοφορίες. 29 υπέρ, καμία ψήφος κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στην ε, εισηγητριά μας. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Και δίνω το λόγο για το σημείο 13. Α, όχι. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, διορθώνει η Πρόεδρος. Πρώτα θα εξετάσουμε το σημείο για το οποίο είναι εισηγητής ο κύριος Φρεντερίκ Νταρντάν που αναβάλαμε για μετά την ψηφοφορία. Είναι τα σημεία 4 και 5 στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για το πακέτο σιδηροδρομικών μεταφορών. Εδώ έχει ζητηθεί γνωμοδότηση από εμά για δύο κείμενα. Το ένα έχει να κάνει με την τροποποίηση του κανονισμού 1370-2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών συνδρομικών μεταφορών και πρόκειται και για την τροποποίηση οδηγίας 2012-34 της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκού Συνδρομικού Χώρου όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών συνδρομικών επιβατικών μεταφορών και την διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής. Παρακαλώ κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε τις συμβιβαστικές τροπολογίες σχετικά με τις δύο αυτές εκθέσεις. Παρακαλώ κύριε Ταρντά. Σας ευχαριστώ, θα είμαι σχετικά σύντομος. Τρία σημεία θέλω να τονίσω. Να σας υπενθυμίσω καταρχήν την κατεύθυνση που πήρε το σχέδιο έκθεσης και επίσης στην κατεύθυνση των τροπολογιών που κατατέθηκαν. Η δική μου προσέγγιση είναι να πω ότι δεν πρέπει να κάνουμε χωρίς ε, έλεγχο μία απελευθέρωση χωρίς να εξασφαλίσουμε ότι η αλλαγή αυτή των δομών θα αυξήσει την προσβασιμότητα για τους επιβάτες και την ασφάλεια των μεταφορών, επίσης ότι πρέπει να προστατεύσουμε και τους εργαζομένους όταν υπάρχουν τέτοιου είδους αλλαγές στις δομές, παραχωρήσεις κτλ. Ε, δεδομένης τώρα της ε, γενικής σύγκλησης απόψεων μαζί με τους συναδέλφους μου του ΕΛΚ και σε μεγάλο βαθμό με τους πρασίνους σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, εγώ έχω προτείνει κάποιες συμβαστικές τροπολογίες στο βαθμό που υπήρχε κάποια δυνατότητα Υπάρχουν έξι τροπολογίες συμβασμού για την οδηγία που έχω καταθέσει και αρκετές ακόμα για τον κανονισμό. Επί τη βάση των επαφών που είχα μέχρι σήμερα, οι φιλελεύθεροι παραμένουν στη δική τους ε, γραμμή η οποία απέχει αρκετά από αυτή που παρουσίασα προηγουμένως. Πιστεύω λοιπόν ότι ο αρμόδιος της ε, Σκιώδης θα λάβει το λόγο σχετικά και ξέρω ότι δεν πρόκειται να με υποστήριξει ιδιαίτερα για τα θέματα αυτά και επειδή βάσει των επαφών που έχουμε κάνει στο παρελθόν ξέρω ότι υπάρχουν από τους πρασίνους κάποιες αιτήσει για διαφοροποίησεις και τροποποιήσεις στο κείμενο ώστε να μπορέσουμε σήμερα ή αύριο το πρωί τουλάχιστον να καταλήξουμε σε οριστικές συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ. Ποιος θέλει το λόγο? Κύριε Μπακ. Ο Ζος Μπαχ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ. Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου και εγώ να πω ότι όσον αφορά την εισαγωγή και τις παρατηρήσεις για το θέμα της απελευθέρωσης των συνδρόμων, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο συγητής και θέλω επίσης και να τον συγχαρώ ουσιαστικά για τις δύο εκθέσεις του, γιατί δύο είναι οι εκθέσεις και επίσης και να τον συγχαρώ και για τους συμβασμούς που επέτυχε. Συμφωνούμε, δεχόμαστε αυτούς τους συμβασμούς, έτσι κι αλλιώς ο συμβασμός H κατέπεσε, ο M για μένα είναι εντάξει και όσον αφορά τον συμβασμό G τον στηρίζουμε αυτόν ανεπιφύλακτα. Κατ' ουσίαν δηλαδή δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Εγώ θεωρώ ότι πράγματι εργαζόμεθα προς το όφελος των εργαζομένων των συνδρόμων και η έκθεση την οποία θα εκπονήσουμε είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπενιόν και, και μετά η Ελίζαμπεθ Σρέτερ, ο Φιλ, Μπενιόν, Φιλ Μπενιόν. Χωρίς μικρόφωνο ο μιλητής, δυστυχώς. Έχει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα ο μιλητής. He's obviously, he's, he's obviously taken the microphone with him που έφυγε πήρε μαζί του και το μικρόφωνο. Δυστυχώς ο κύριος Ντεμπάκερ ε, δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, αλλά εγώ δούλεψα στην Επιτροπή Μεταφορών για αυτή τη δέσμη μέτρων από κοινού σε συνεργασία με τον κύριο Ντεμπάκερ. Θέλω να πω το εξή ότι πήραμε κάποιες σημαντικές προτάσεις από τον εισηγητή, αλλά έπρεπε να γίνουν κάποιες και οδόν, δεν έλαβαν αυτές χώρα και δεν ελήφθησαν υπόψη οι τροπολογίες ε, στο συμβασμό. Νομίζω αυτό το είπε ήδη ο εισηγητής. Κατόπιν του δεν θα μπορέσουμε να στηρίξουμε όλες τις τροπολογίες, θα στηρίξουμε κάποιες εξ αυτών. Κυρίως όσον αφορά τον κανονισμό. Νομίζω εκεί πραγματικά έχουμε μεγάλη δυσκολία. Οι συμβαστικές προτάσεις B, E, F, G, I, K, M και N όσον αφορά αυτές τις συμβαστικές και το τελευταίο κομμάτι της συμβαστικής π, αυτές δεν μπορούμε να τις ε, στηρίξουμε. Σε επίπεδο κυβέρνησης θέλουμε να πούμε μάλλον διακυβέρνησης. Εκεί θέλουμε να πούμε ότι οι συμβαστικές προτάσεις ακολουθούν τελείως αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που πιστεύουμε εμείς. Κατόπιν τούτου και αυτές για τη διακυβέρνηση δεν θα μπορέσουμε να τις στηρίξουμε. Να πω και κάτι άλλο ε, σχετικά με το ότι λυπούμεθα για το ότι οι συμβαστικές προτάσεις ακολουθούν τελείως διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν που ακολουθεί η Ευρώπη εδώ και χρόνια και από αυτήν που προτείνει η Επιτροπή. Γίνονται πάρα πολλέ συζητήσει σχετικά στην Επιτροπή Μεταφορών το άνοιγμα των αγορών και η διακυβέρνηση μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές επιπτώσεις γενικά για την αγορά των σιδηροδρόμων αλλά και για τους εργαζόμενους στον τομέα των σιδηροδρόμων. Η εμπειρία από το ΕΒ και τη Σουηδία από αυτά τα δύο κρατημέλη που ακολούθησαν αυτή την κατεύθυνση με τις δικές τους τις συνδρομικές υπηρεσίες αποδεικνύουν αυτό τον ισχυρισμό. Γιατί σε αυτές τις δύο χώρες αυξήθηκε η απασχόληση στον τομέα των σιδηροδρόμων. Το να διατηρήσει κανείς το ισχύον καθεστώς, αυτό είναι ζημιογόνο. Οι επιβάτες ε, και οι οικονομίες των κρατών στη τελική ανάλυση θα καταστούν θύματα ενδεχομένως αυτής της εξέλιξης. Η κυρία Σλούτα έχει το λόγο. Σρόντερ, με συγχωρείτε. Εγώ λοιπόν θα εξετάσω ξεχωριστά ε, όλα αυτά τα θέματα. Καταρχήν, πρόκειται για την οδηγία. Όσον αφορά την οδηγία, εμείς είχαμε παρακαλέσει στη συμβαστική D αυτό να μην εμφανίζεται ως συμβιβασμό, αλλά να έχει τη μορφή δύο διαφορετικών τροπολογιών. Διότι δεν πρόκειται για συμβασμό. Οι ε, τροπολογίες ε, απλά αναφέρονται με αλουχία, η μία μετά την άλλη. Και εγώ θα προτιμούσα να γίνει ψηφοφορία επί των τροπολογιών, ε, τη στιγμή μάλιστα που η προστίκη του εισηγητή σε αυτό το άρθρο είναι κατ' ουσίαν μία προστίκη. Άρα δηλαδή μπορεί να ψηφιστεί εν είδη Ενώ η δική μας τροπολογία είναι κανονική τροπολογία. Εγώ είχα καταλάβει ότι ο εισηγητής συμφωνεί με τη δική μας την τροπολογία. Δυστυχώς όμως μετά από αυτή την πρόταση που καταθέσαμε, δηλαδή να ψηφίσουμε κανονικά τροπολογίες και μετά την προστίκη με τη μορφή προστίκης, όσον αφορά αυτή τη θέση μας, δυστυχώς δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά στον κανονισμό. Στον κανονισμό είχαμε καταθέσει κάποιες προτάσεις. Παραδείγματος χάρη, πώς είναι δυνατόν στις συμβαστικές προτάσεις να βελτιωθούν, να συμπεριληφθούν βελτιωμένες οι τροπολογίες μας. Διότι το κείμενο που μας κατέθεσε ο συγητής δεν κατιστά σαφές κατά πόσον οι τροπολογίες μας πράγματι περιλαμβάνονται βελτιωμένες ή όχι. Και αυτό αφορά κυρίως την τροπολογία υπαριθμών Β. Εκεί είχαμε καταθέσει ε, πρόταση βελτίωσης. Ο εισηγητής δεν αντέδρασε σε αυτό. Ίσως μπορεί να αντιδράσει βέβαια τώρα. Όσον αφορά τη συμβαστική G, Εκεί υπάρχει ένα θέμα το οποίο όμως ε, δεν στηρίζουμε. Πρόκειται για κάτι που αναφέρεται στην αρχή. Εμείς ε, θα θέλαμε να υπάρχει η πρωτότυπη διατύπωση. Ο συγητής είπε ότι ε, θα ανταποκριθεί σε αυτό. Αλλά μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε ποια είναι η θέση του επ' αυτού. Έχουμε μόνο την αντίδραση του συναδέλφου Μπαχ, ο οποίος, όπως το είπε έτσι πολύ λεπτά, συμφωνεί με τις δικές μας τις τροπολογίες. Και πραγματικά με μεγάλη περιέργεια περιμένω να δω τι θα πει επ' αυτόν ο εισηγητής. Για την Κομισιόν. Κυρία Προύτ, θέλει να λάβει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, κυρία Πρόεδρε. βάσει των εμπειριών που είχαμε στα διάφορα κράτη-μέλη, η Κομισιόν επέλεξε μια εξισορροπημένη και βαθμιαία διαδικασία για το να ανοίξουν οι αγορές επιβατών στον ανταγωνισμό. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει τη διατήρηση των προνομίων που έχουν τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των υποχρεώσεων για τις δημόσιες υπηρεσίες και θέλουν να αποτρέψουν την επιλεκτική συμπεριφορά στα θέματα αυτά τα, κράτη, τα μελη πρέπει να εξασφαλίσουν την καλή κατάρτιση του προσωπικού στους σιδηροδρομικούς φορείς και με τη διαδικασία δημοσίων διαδικασιών διαγωνισμών μπορεί να εξασφαλιστεί ένα μεγάλο επίπεδο εξοικονομήσεων. Οι κοινωνικές επιπτώσεις φυσικά είναι ένα θέμα που απασχολεί την Επιτροπή σας και ο συγητής έχει κάνει προτάσεις για βελτίωση σε ορισμένα σημεία της πρότασης της Κομισιόν για την Οδηγία 212-34, 2012-34, 34 παραγωγή καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών υποδομών ή για τον ε, κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές ε, διαπραγματεύσεις, όπως οι τροπολογίες 4 και 5, συμμετοχή των κοινωνικών εστέρων στην Επιτροπή <clears throat> Συντονισμού, τροπολογία 11 και επίσης και για άλλες τροπολογίες που στην διακατεύθυνση, όπως η 61 και 69 της κυρία Σρέτερ ή 66 και 67 από τον κύριο Λούντβικ Σον. Η Κομισιόν χαιρετίζει όλες τις τροπολογίες οι οποίες βελτιώνουν το πλαίσιο για ένα πιο δυναμικό χώρο αγοράς για τους ιδιοδρομικούς φορείς και για ανεξαρτησία των διαχειριστών υποδομών, όπως είναι η τροπολογία 46 και οι τροπολογίες 50 με 53 και 57 η τροπολογία επίσης 54, 58 και η 70. Οι τροπολογίες όμως που θέλουν να αποδυναμώσουν ή να διαγράψουν τις πρόνοιες της πρότασης Κομισιόν για κάθετη ολοκλήρωση των δομών μας φαίνονται προβληματικές. Αυτό εσύ για τις τροπολογίες 11, 12, 13, 49 και ιδιαίτερα για την 56 του εισηγητού. Οι τροπολογίες αυτές αφορούν σημαντικά και ουσιαστικά στοιχεία της πρότασής μας, τον ορισμό των ε, κάθετα και χωρισμένων δομών, την ανάγκη για διαφάνεια, τους κανόνες για τις διαχειριστικές τομές σύγκρουση συμφερόντων, μηχανισμούς επαλήθευσης, που όλα αυτά είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί ισότητα ανταγωνισμού για όλους τους εμπλεκόμενους. Έχουμε επιφυλάξει επίσης τις τροπολογίες που επιβάλλουν τη δημιουργία κοινών συστημάτων πληροφόρησης και έκδοσης εισιτηρίων εν ώψη της ε, ενσωμάτωσης των αγορών και της διατήρησης της εμπορικής ελευθερίας των σιδηροδομικών φορέων και επίσης για την επίτευξη κάποιας ισορροπίας στα νέα συμβόλαια και τις νέες συμβάσεις που θα δημιουργηθούν. Επίσης οι προτάσεις που αφορούν ορισμένα άρθρα που έχουν να κάνουν με τη δοκιμασία οικονομικής ισορροπίας και την ανάγκη να σέβονται τις συλλογικές συμβάσεις της Ιδροδομικής Φορής καθώς και τις ανάγκες αναφορών από την Κομισιόν για την ανάπτυξη της εργασιακής αγοράς. Η Κομισιόν μπορεί να δεχτεί καταρχήν αυτές τις τροπολογίες. Αν μπορώ να πω κάτι και για τον κανονισμό σε σχέση με τις συμβασικές τροπολογίες για τον κανονισμό 1370 η Κομισιόν συμφωνεί με την ενίσχυση των διαδικαστικών μέτρων για διαφάνεια και χαιρετίζει τις τροπολογίες συμβασμού J και L που θέλουν να διευρύνουν τη διαβούλευση για τα δημόσια σχέδια μεταφορών με σιδηροδρόμους και τις δημόσιες υποχρέωσεις υπηρεσιών ώστε να καλύπτουν και άτομα που είναι ηλικιωμένα ή έχουν αναπηρίες. Η Κομισιόν χαιρετίζει επίσης τη συμβαστική τροπολογία O η οποία θεσπίζει και μια αρχή αμοιβαιότητα για τι εταιρείε που ελέγχονται από φορείς σε τρίτε χώρε. <clears throat> το τμήμα τη τροπολογία συμβασμού Q που προτείνει στην ετήσια έκθεση να περιλαμβάνεται και από τι αρμόδιες αρχέ μια αξιολόγηση τη απόδοση των επιχειρήσεων σιδηροδρόμου και τη ε, πληρότητά του είναι επίση καλόδεκτη. Αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε δημιουργία πρόσθετου διοικητικού άκθους για τις εθνικές αρχές η Κομισιόν δεν βλέπει θετικά τις τροπολογίες M και N, την, ε, την επιβολή μεταφοράς προσωπικού παραδείγματος χάρη και επίσης τα, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα τα οποία θέλουν να επιβάλλουν. Γιατί είναι ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά των συνδρομικών αγορών και της εργασιακής αγοράς τους στα διάφορα κράτη-μέλη. Βάσει της αρχής επικουρικότητας θα πρέπει να επαφείται στις εθνικές και περιφερειακές αρχές να κρίνουν και να αποφασίσουν για τα μέτρα προστασίας του προσωπικού. Η Κομισιόν δεν θέλει να περιορίσει το επίπεδο ελιγμών των κρατών μελών εάν θέλουν να δώσουν τα κράτη-μέλη διαφορετικά τμήματα της αγοράς σε διαφορετικές επιχειρήσεις και για να εξασφαλίσουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, όπως λέει η Συμβαστική Τροπολογία Π. Τέλος, η Κομισιόν θεωρεί το δεύτερο τμήμα της Τροπολογίας Συμβασμού Q, που ζητά από την Κομισιόν να κάνει μια συμπίληση και σύνοψη εκατοντάδων εκθέσεων από εθνικές και περιφερειακές αρχές και να μεταφράσει όλα αυτά τα ε, επίτομα έγγραφα, θα, θα σημαίνει ένα τεράστιο διοικητικό άχθος που δεν θα οδηγήσει σε θετικούς καρπούς. Ευχαριστώ μου δώσατε το λόγο. Πολύ καλά. Νομίζω ότι τα μέλη της Επιτροπής χαίρονται πάρα πολύ που ακούσαν την άποψη της DG Move ε, που φαντάζομαι ότι την ίδια απόψη έχει και η Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση. Χαιρόμαστε για το γεγονός ότι η Κομισιόν μας έχει δώσει την άποψή σας μέσα στα πλαίσια αυτά και φυσικά ελπίζω ότι θα δώσει τα στοιχεία αυτή και στην Επιτροπή Μεταφορών και θα ήθελα να δώσω και πάλι το λόγο στον εισηγητή για να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους όσοι πήραν το λόγο και για τη συνεργασία. Τώρα, όσον αφορά το είπε ο κύριος Μπενιό, ο οποίος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη συνεδρίαση σκιωδών ε, ουσιαστικά έχει οργανωθεί, αλλά μετά χρειάστηκε να ακυρωθεί γιατί δεν ήταν ε, διαθέσιμοι όλοι οι σκιώδε. Και μετά με mail ανταλλάξαμε απόψεις και έτσι νομίζω ότι προχωρήσαμε και ξέραμε τι υποστηρίζει ποιο σε σχέση με τις συμβαστικέ τροπολογίες. Ε, δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επί της ουσίας. Είναι προφανές αυτό σήμερα. Για τις αντιδράσεις της κυρίας Ρέντερ τώρα. Όσον αφορά την οδηγία, συμφωνώ με την παρατήρησή της και με την πρότασή της να αποσύρουμε τον συμβιβασμό αυτό και να έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία, χωριστά μάλλον, τις τροπολογίες που συμπεριλαμβάνονται στο συμβασμό Δέλτα. Όσον αφορά τον κανονισμό, εδώ έχετε τρεις προτάσεις. Υπάρχει πρόταση που μπορούμε να συζητήσουμε ακόμα περισσότερο μεταξύ μας για να καταλήξουμε τελικά τι θα κάνουμε τις αλλαγές που προτείνετε. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε πάντως μέσα στις επόμενες ώρες να βρούμε μια συμφωνία μεταξύ μας και έτσι να έχουμε και ένα τελικό κείμενο συμβαστικής τροπολογίας. Έρχομαι τώρα στις άλλες τροπολογίες, ή μάλλον στα άλλα σχόλια και παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ για την λεπτομερή αυτή ανάλυση που κάνετε όσον αφορά το έργο μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ για το θέμα αυτό. Τελειώσαμε. Θα το ψηφίσουμε στις 18 Νοεμβρίου. Η Επιτροπή Μεταφορών θα ψηφίσει στις 26 Νοεμβρίου. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο 13 στην ημερήσια διάταξη. Το λόγο έχει μια κρίσταλο που θα μας ενημερώσει για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βοήθειας προς τους Απόρους. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Συμβούλιο ε, συμφώνησε ε, στο πλαίσιο της ε, τριμερούς ε, συζήτησης που έλαβε χώρα που ξεκίνησε στις 16 Οκτωβρίου. Έκτοτε βέβαια είχαμε τρεις συναντήσεις, ε, τριμερείς ε, συναντήσεις και τελικά βρεθήκαμε σε τεράστια πίεση χρόνου. Όσον αφορά τώρα τις προτάσεις που κατατέθηκαν, θα γνωρίζετε ότι υπήρχε μια αποκλείουσα, μια μειοψηφία που μπλοκάριζε τη λήψη αποφάσεων βέβαια σε σχέση με το πρόγραμμα και σε σχέση με την ψηφιστική βοήθεια, την διανομή της. Το Συμβούλιο επανήλθε με νέες προτάσεις και αυτό το οφείλει το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μεγάλο βαθμό. Κατορθώσαμε να διασφαλίσουμε άλλο ένα δις ευρώ. Ε, έτσι λοιπόν ο προεπλογισμός αυξήθηκε σε 3,5 δις ευρώ. Η συμφωνία του Συμβουλίου προτείνει να αλλάξει η πρόταση με διάφορους τρόπους. Καταρχήν προτείνεται να υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα το οποίο θα περιφέρει μεγαλύτερο εύρος εφαρμογής του τρέχοντος προγράμματος, δηλαδή να περιλαμβάνεται και το θέμα του, της κατάργησης κοινωνικού αποκλεισμού, μέτρα που ε, προβλέπουν την ε, κατάργηση, όπως σας είπα, του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως είχε προβλεφθεί και στην αρχική πρόταση. Όσον αφορά της, ε, τη διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της οποίας ηγείται η πρόεδρος, η κυρία Μπερέζ, εγώ και οι σκιώδεις εισηγητές εξετάσαμε τις προτάσεις του Συμβουλίου Βέβαια εμείς είχαμε τις δικές μας ανησυχίες για την παράταση και πολλές από τις ανησυχίες μας είχαν σχέση με τα θέματα τα οποία συζητήσαμε όταν συζητήθηκε αυτή η πρόταση στην Ολομέλεια και παλαιότερα στην Επιτροπή. Δηλαδή τα κονδύλια για τους άπορους ε, να καταλήγουν πράγματι σε αυτούς και με τον τρόπο αυτό να αποφεύγουμε οποιαδήποτε επικάλυψη με προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου. Επίσης, το Συμβούλιο πρότεινε κονδύλια από τον προπλογισμό λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα έξτρα ένα δις ευρώ που θα κατατεθούν, που θα εκταμιευτούν και κατέληξε σε μία πρόταση για ε, κονδύλια από το Ταμείο το ΦΕΑΝΤ που προβλέπεται για τους άπορους. Έτσι λοιπόν να έχουμε ένα ελάχιστο ποσό 3,5 δις ευρώ ανακράτος μέλος. Υπήρξαν αρκετά θέματα όπου το κείμενο του Συμβουλίου αποκλίνει βέβαια από αυτό που είχε προτείνει το Κοινοβούλιο, κυρίως σε σχέση με την αρχή της εταιρική σχέσης. Εμείς επιθυμούμε να συμμετέχουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τόσο στο σχεδιασμό, όσο στην εφαρμογή, όσο και στην αξιολόγηση του προγράμματος ΦΕΑΝΤ. Επίσης, εμείς θελήσαμε να βελτιώσουμε τις προτάσεις του Συμβουλίου, κυρίως όσον αφορά την τοπική αλυσίδα εφοδιασμού, επίσης όσον αφορά την υγιεινή διατροφή και την υγιεινή διαμονή. Θελήσαμε να βρούμε κάποιες μορφές συνεργασίας σε αυτούς τους τομείς. Είχαμε λοιπόν κάποιες συζητήσεις και συζητήσεις αυτές έγιναν με το Συμβούλιο. Καταλήξαμε στο ότι μπορούμε τελικά να δεχτούμε την διευρυμένη εφαρμογή υπό την προϋπόθεση ότι η νέα αυτή πρόταση για το μη αποκλεισμό αφορά τους πραγματικά άπορους και δεν θα υπάρχει επικάλυψη με το ESF το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Επίσης, ε, επιμένουμε το θέμα της ε, συνεργασίας ε, με κοινωνικές πολιτικές για την αλυσίδα εφοδιασμού, για την υγιεινή διατροφή και όλα τα συναφή, αυτά θα ληφθούν υπόψη. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε μία σειρά τροπολογιών έτσι ώστε να διασφαλίσουμε αυτές οι αρχές για τις οποίες εργαστήκαμε τόσο σκληρά, αυτές πράγματι τελικά να διατηρηθούν. Ένα άλλο θέμα το οποίο προέκυψε σε σχέση με τις ε, προτάσεις του Συμβουλίου είναι τα θέματα που αφορούν στα κοινωνικά παντοπολία. Αυτά ε, νομίζω ε, αφορούν σε όλα τα κράτη-μέλη, έχουν σχέση με την επισητιστική βοήθεια, τη βοήθεια παροχής τροφίμων. Ένα άλλο θέμα αφορά στα μεταβατικά μέτρα. Όλοι μας ανησυχούμε διότι επιθυμούμε το πρόγραμμα αυτό να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν και χωρίς καμία καθυστέρηση. Γι' αυτό λοιπόν επιθυμούμε διακαώς να υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις που θα τεθούν σε ισχύ έτσι ώστε το πρόγραμμα πράγματι να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και τα κράτη-μέλη και οργανώσεις ε, που συνεργάζονται με τους πραγματικά άπορους να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη χρηματοδότηση από την 1η Ιανουαρίου. Να μην δηλαδή τιμωρηθούν ε, κατά κάποιον τρόπο. Επί της ουσίας, σας είπα, είχαμε τρεις ε, τριμερείς ε, συζητήσεις, σημειώσαμε πρόοδο, ε, συστήθηκαν αρκετές ομάδες εργασίας τεχνικής φύσεως επί του θέματος και προβλέπουν και άλλες τρει τριμερείς συζητήσει. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για τη συνεισφορά τους. Νομίζω ότι όλοι δούλεψαν σκληρά για να επιτευχθεί η συμφωνία. Συνεργάστηκαν όλοι οι σκιώδεις εισηγητές για την κατάθεση των προτάσεων και α μην ξεχνάμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ε, διασφαλίσουμε μια συμφωνία. Η τελευταία τελευταία τριμερή ε, συζήτηση θα λάβει χώρα στις 28 Νοεμβρίου και εκεί θα είναι η τελευταία πρόκληση και ευκαιρία που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε. Ποιος θέλει το λόγο, η κυρία Σαρτιέ, ο Σαρτιέ και μετά και εγώ να έχω να πω δύο λόγια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα και ευχαριστώ ειλικρινά τη συνάδελφο Κοστέλο για όλη τη δουλειά που έχει κάνει για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και για τη συμμετοχή της στους τριμερείς διαλόγους. Η Καστέλο το είπε και ίδια ότι υπάρχει ένα σημείο που για μας είναι ουσιώδης και είναι αυτό των κοινωνικών παντοπολίων. Έτσι όπως διατυπώνεται σήμερα το κείμενο, αποκλεί πλήρως χρηματοδοτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην διανομή των τροφίμων. Ενώ τα κοινωνικά αυτά παντοπολία ζητούν ένα πολύ χαμηλό ποσό και από ό,τι ξέρω, από τις επαφές που είχα, μου αποδεικνύουν ότι τελικά το κοινό που έρχεται, οι πελάτες, είναι τόσο διαφορετική μεταξύ τους ακριβώς γιατί το μικρό αυτό ποσό συνεισφοράς τους επιτρέπει να μην δέχονται τελικά ελεημοσύνη, δέχονται μια βοήθεια από το Ταμείο για τους Απόρους, αλλά είναι καλό να νιώθει κανείς την ανάγκη για αξιοπρέπεια. Μερικές φορές είναι νέοι φοιτητέ, οι οποίοι δεν θέλουν τα πάντα δωρεάν, αλλά θέλουν να συνεισφέρουν κάπως. Οπότε, έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, έτσι δηλαδή όπως είναι διατυπωμένο σήμερα το κείμενο, η δυνατότητα αυτή αποκλείεται. Αυτό κατά τη γνώμη μου θέτει σε κίνδυνο τα ίδια τα κοινωνικά πατοπολία, τα οποία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό λοιπόν ήθελα να πω πέρα από τα μέτρα εφαρμογής, γι' αυτό ήθελα να μιλήσω όλος ιδιαίτερος και ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ θέλω να μιλήσω για αυτό το σημείο, το είπε και η ότι άνοιξε η συζήτηση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για αυτό το θέμα και είπαμε ότι θα μεταφέραμε στο Συμβούλιο μία πρόταση η οποία να βασίζεται σε τρία σενάρια. Πρώτον, τροπολογία όπως την ψήφισε η Επιτροπή Γεωργίας και η Επιτροπή Προϋπολογισμών, αλλά που δεν συμφώνησε δικιά μας η Επιτροπή ώστε να προβλέψουμε πως σε μερικές περιπτώσεις τα προϊόντα που διανέμονται μέσω του προγράμματος αυτού να χρεώνονται 10% της ε, αξίας τους. Δεύτερη επιλογή είναι απλά να χρησιμοποιήσουμε την διάταξη που υπάρχει σήμερα για το Ταμείο στο πρόγραμμα μάλλον έτσι όπως έχει σήμερα. Κάτι το οποίο βέβαια έρχεται σε αντίφαση με αυτό που λέει η Κομισιόν, γιατί η Κομισιόν μας λέει ότι είναι δύσκολο να έχουμε δύο διαφορετικούς λογαριασμούς ανάλογα με το κατά πόσο η τιμή του προϊόντος ε, φέρνει έσοδα ή όχι. Από την άλλη όμως η Κομισιόν συμφώνησε με το Συμβούλιο όταν αποφάσισε για ένα παράλληλο πρόγραμμα λειτουργικό. Οπότε έτσι γίνεται κάποια επικάλυψη, ενώ θα μπορούσαμε να καλυφθούμε από αυτή την νομοθεσία. Εγώ δεν καταλαβαίνω το επιχείρημα της Εκτελεστικής Επιτροπής. Και το τρίτο σενάριο που προτείνω, σε συμφωνία με την εισηγήτρια, είναι στα πλαίσια του άρθρου 7 του κειμένου να προβλέψουμε εξαίρεση από τις χώρες μέλη στο θέμα της δωρεάν διανομής προϊόντων που περιλαμβάνονται στο λειτουργικό πρόγραμμα Food and Material Assistance. Η διαπραγματευτική ομάδα στη βάση αυτή θα διατυπώσει μια πρόταση η οποία θα πάει στο Συμβούλιο πριν από την τριμερή συνάντηση που θα έχουμε, τον τριμερή διάλογο. Άλλος κανείς, δεν βλέπω να θέλει κανένας άλλος το λόγο, η συγκίτρια λοιπόν και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά με το Συμβούλιο και την Κομισιόν σε σχέση με το πρόγραμμα αυτά, αυτό. Είναι σημαντικό όμως να εξασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια που θα πάρουμε για το πρόγραμμα αυτό θα ανταποκριθούν στις ανάγκες των δικαιούχων. Πολλές φορές μιλάμε για άτομα τα οποία είναι περιθωρικοποιημένα και αντιμετωπίζουν προβλήματα οξίας ένδυας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεχάσουν την αξιοπρέπειά τους οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν. Προσπαθούμε να καταλήξουμε λοιπόν με ένα σύνολο εναλλακτικών προτάσεων που θα μπορέσουμε να οδηγήσουν σε μια ικανοποιητική επίλυση αυτού του προβλήματος και το Συμβούλιο και η Κομισιόν, όπως είπε και η Πρόεδρός μας, τόνισαν ότι υπάρχουν ακόμα κάποια προσκόμματα Κατανοούμε όμως ότι μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και ακριβώς αυτός είναι ο στόχος μας να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ενώπιών μας. Αλλά θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι έχουμε μεγάλη πίεση χρόνου και είναι σημαντικό να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει συμφωνία για αυτό το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε καμιά δυνατότητα τριγωνικών διαλόγων το Δεκέμβριο και θέλουμε όπως και οι αρμόδιοι φορείς που υποστηρίζουν τα άτομα αυτά που εξαρτώνται από αυτή την μορφή αρρωγής, θέλουμε πάρα πολύ να προσπαθήσουμε το ταχύτερο δυνατό να εξασφαλίσουμε την έγκριση αυτού του προγράμματος. Ευχαριστώ και πάλι όλους τους συναδέλφους για την ενθάρρυνσή τους και τη συνεργασία τους και είμαι σίγουρη ότι με την συνέχιση αυτής της συνεργασίας θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας και να κλείσουμε ικανοποιητικά το θέμα αυτό μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπέρας χρειάστηκε να απουσιάσει για λίγο. Θα συνεχίσω στα πορτογαλικά. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 14. Αλλά επειδή και η πρόεδρος μας είναι εκτός αίθουσες, εγώ θα πρότεινα να περάσουμε στο σημείο 15 για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και επίσης σε σχέση με τα θέματα δημοσιονομικής διαφάνειας των λιμένων. Ο εισηγητής για το θέμα αυτό είναι ο Φιλίπ Τεμπάκερ από τους φιλελεύθερους, ο οποίος δεν είναι παρόν από ό,τι γνωρίζω. και προβλέπεται να τον αντικαταστήσει για την παρουσίαση αυτής της ε, γνωμοδότησης ο κύριος Μπένιον. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, είπαμε και προηγουμένως ότι ο Ντεμπάκε ε, δεν παρίσταται και έχω έρθει εγώ για να παρουσιάσω το σχέδιο της εκθεσής του για πρώτες κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση ε, πλαισίου για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και την διαφάνεια των λιμένων. Η κύρια επιτροπή είναι η Επιτροπή Μεταφορών, η τα ε, λιμάνια απασχολούν πάνω από 3 εκατομμύρια άτομα ε, άμεσα ή έμεσα. Έχουμε λοιπόν ε, και τα λιμάνια τα οποία συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις όμορες περιοχές. Πρέπει να υπάρξει νομοθεσία γιατί αυτή τη στιγμή τα μέτρα που ισχύουν απλά δημιουργούν νομική ανασφάλεια. Έχουμε λοιπόν μια πρόκληση για την επίτευξη κοινωνικής προστασίας αφενός και ε, οικονομικής βιωσιμότητας απετέρου να στηρίξουμε τους παρόχους υπηρεσιών και τις υπηρεσίες των λιμένων. Η γνωμοδότηση είναι αρκετά ευσύνοπτη προτείνεται να υπάρξει ελευθερία στην παροχή υπηρεσιών από πλευρά λιμένων, να ανοίξει η αγορά, γιατί αυτό θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, θα υπάρχει καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Η νομική ασφάλεια για τα λιμάνια επίσης θα πειράσει και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Ο Φιλίπ αναγνωρίζει ότι όταν οι ε, εργαζόμενοι δουλεύουν στα λιμάνια αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να διασφαλιστεί η σωματική του ακαιρεότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και στηρίζει την άποψη ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν θα επηρεάσει την ε, κοινωνική κατάσταση των εργαζομένων. Όσον αφορά του εργαζόμενου, ε, ο Φιλίπ προτείνει τον διάλογο, πρέπει να υπάρξει ε, κάποια συμφωνία και στα εδάφια που ακολουθούν καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένη συμφωνία. Τονίζει επίσης ότι πρέπει να συμπληρωθεί ο κοινωνικός διάλογος, ε, σίγουρα όχι να αντικατασταθεί. Προσβλέπει στο να υπάρχει ε, συνεχής επαφή με τους σκιωθηγητές και ευχαριστεί για την ε, συνεργασία έτσι ώστε να υπάρξει μια ικανοποιητική γνωμοδότηση. Ο κύριος Μπαχ τώρα έχει το λόγο. Σας σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ε, πράγματι δεν έχουμε προβλήματα με την κατεύθυνση που ακολουθεί αυτή η πρόταση της Επιτροπής. Ε, σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ με αυτά που είπε ο Σνάλφος Μπένγκεμιν και συμφωνώ ε, και με αυτά που προτείνει ο κύριος Ντεμπάκελ ε, νομίζω λοιπόν ότι οι οικονομικές ε, προκλήσεις, ε, η ασφάλεια των εργαζομένων, οι συνθήκες εργασίας, όλα αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και εξίσου σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η Επιτροπή έκανε δύο αποτυχημένες προσπάθειες και έμαθε εξ αυτών. Έτσι λοιπόν τώρα πλέον η Επιτροπή το όλο θέμα ε, των κοινωνικών και εργασιακών διατάξεων δεν το περιλαμβάνει σε αυτή την πρόταση. Στον, ε, τα θέματα αυτά θα εξεταστούν περισσότερο στον ειδικό τομεακό διάλογο και αυτό το χαιρετίζω. Ε, όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο, πολύ συχνά έχει προκύψει οδηγία από κοινωνικό διάλογο μετά από συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και αυτό το βρίσκω ιδιαίτερα θετικό. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή δεν τίθεται αυτό το θέμα για μας. Ο συνάδελφος Μπένιαμιν μίλησε για το 2016. Νομίζω λοιπόν ότι αν οι κοινωνικοί εταίροι δεν καταλήξουν, τότε θα πρέπει να επιληφθούμε και πάλι του θέματος αυτού. Όμως δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Εγώ εναποθέτω τις ελπίδες μου στον κοινωνικό διάλογο. Όσον αφορά το εκτιμώντας 10, νομίζω ότι πρέπει να το δουλέψουμε λιγάκι το εδάφιο αυτό και εγώ προσωπικά ε, θα προσπαθήσω αυτό το άρθρο, το άρθρο υπαριθμών 10, να λάβει μια πιο έντονη διατύπωση. Αυτά είχα να σας πω προς το παρόν και βεβαίως προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σουέτερ, η οποία είναι αντιπρόεδρος στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ, λέει κυρία Σουέτερ. Ανεφέρθη ήδη από τον κύριο Μπαχ ότι είχαμε δύο ήδη γύρους συζητήσεων για, την, ε, για το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, Νομίζω ότι το θέμα του κοινωνικού διαλόγου θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην προβληματική μας, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα, το κατά πόσο αυτό μπορέσει να γίνει. Υπάρχει βέβαια το πρόβλημα ότι χρειάζεται υψηλό ποσοστό <clears throat> στις, ε, στην ψηφοφορία, χρειαστεί ειδική πλειοψηφία για να περάσει κάτι τέτοιο. Το κατά πόσο λοιπόν μπορέσουν να γίνουν, να εγγραφούν όλα αυτά τα σημεία στην ε, έκθεση αυτή λοιπόν για μένα είναι κάτι το οποίο αφορά ιδιαίτερα την προστασία των εργαζομένων, την ασφάλειά τους και αυτό είναι ένα θέμα ευρύτερης διάστασης. Πιστεύω λοιπόν ότι στο έγγραφο αυτό να εξασφαλίσουμε τη συμπερίληψή του και πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες προσπάθειες. Η Κομισιόν δεν μπορεί να συγχαίει τώρα αυτό το θέμα με τα προηγούμενα θέματα που αντιμετωπίσαμε προηγουμένως, προτάσεις της Κομισιόν, γιατί δύο φορές απορρίφθηκαν από το Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε όμως μια ιδιαίτερη πλειοψηφία από το Συμβούλιο και εγώ δεν καταλαβαίνω ποια είναι η σύνδεση μεταξύ των δύο αυτών σημείων. Επομένως θα πρέπει να μπει μέσα στον πυρήνα των ε, διατάξεων αυτής της έκθεσης προστασία των εργαζομένων. Ε, ε, Ευχαριστώ κυρία Σρότερ, λέει και η Προεδρεύουσα, δίνω το λόγο. Δίνω το λόγο στον κύριο Θεολογίτη, εξ ονόματος της Κομισιόν. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε και κύριοι. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και να συγχαρώ την Επιτροπή Απασχόλησης για το πολύ καλό έργο που έφεραν πέρας, σε πέρα στην έκθεση αυτή. Πιστεύουμε ότι οι κύριοι στόχοι του κανονισμού μας έχουν γίνει κατανοητοί από την Επιτροπή σας. Πρόκειται για ένα κανονισμό <clears throat> που έχει σαν στόχο να ενισχύσει την θέση των λιμένων και τη θέση του στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφορών. Ενισχύει με τον τρόπο αυτή, αυτή η έκθεση την οικονομική ανάκαμψη και επίσης συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Στην έκθεση αντικτύπου μας έχουμε τονίσει το ότι ένα εκατομμύριο τόνων πρόσθετου φορτίου που μεταφέρεται σημαίνουν 300 θέσει εργασία για καθελημένα. Αυτό δεν είναι η αξιολόγηση της ίδιας Κομισιόν είναι από τα στοιχεία του ΟΣΑ στην έκθεσή του για τους λιμένες και τις πόλεις. Η συνολική ροή από ευρωπαϊκούς λιμένες αυτή τη στιγμή είναι κάτι λιγότερο από 4 δισεκατομμύρια τόνους και ελπίζουμε πιστεύουμε ότι θα υπάρξει σημαντική ανάπτυξη και τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό θέλουμε να δώσουμε στα λιμάνια μια ασφάλεια δικαίωση ό,τι αφορά τις επενδύσεις και ισότητα ανταγωνισμού που είναι μια από τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη στους διάφορους αυτούς τομείς. Αυτή η πρόταση περιέχει μια προσέγγιση εργαλειοθήκης, δεν είναι μια πρόταση η οποία έχει μια ενιαία ε, συνταγή για όλα τα θέματα, Ελπίζω το αναγνωρίζουν αυτό τα μέλη της Επιτροπής σας, ότι η πρόταση αυτή δίδει στις αρχές της λιμενικές και στα κάτι μέλη μια σειρά διαδικασιών με τις οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα όλων των φορέων που εμπλέκονται στους λιμένες και ιδίως Θέλω να υπογραμμίσω ότι με την πρόταση αυτή τα κράτη-μέλη προσκαλούνται να θεσπίσουν υψηλές προδιαγραφές για την κατάρτιση του προσωπικού και να εξασφαλίσουν και τα θέματα ασφάλειας και υγείας που αναφέρθηκαν στις παρεμβάσεις των βουλευτών. Έχουμε προσεκτικά Έχουμε σταθεί προσεκτικοί στο να αποκλείσουμε τα εργασιακά θέματα από την πρότασή μα, εκτό από μια συγκεκριμένη περίπτωση, όταν θέλαμε να εξασφαλίσουμε τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων σε ένα τομέα ο οποίο είναι εν μεταβάση, θα εξασφαλιστούν. Και νομίζω ότι αυτό έχει αναγνωριστεί και από τον εισηγητή στι τροποποιήσει που έχει προτείνει για τι αιτιολογικέ σκέψει και στο εκτελεστικό τμήμα <clears throat> τη πρόταση για την διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων και συγχρόνως μετά από μια μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων με τους εμπλεκομένους έχουμε δημιουργήσει μια επιτροπή κοινωνικού διαλόγου που έχει σαν εγχείρημά της το να εξασφαλίσει τα θέματα της υγείας και της ασφάλειας που είναι πρωταρχική σημασία και να εξασφαλίσει επίσης και τα πρότυπα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχει ξεκινήσει να εργάζεται αυτή η Επιτροπή ήδη θα υπάρξει άλλη μια συνεδρίαση που θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου και πολλές ακόμα το 2014 και θέλουμε με τον τρόπο αυτό να παρακολουθήσουμε το έργο των κοινωνικών εταίρων στις περαιτέρω συζητήσεις τους. Εν κατακλείδη, θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου που έχουν εκφράσει την άποψή τους για το θέμα αυτό. Πρόκειται για μια στάση η οποία είναι υποστηρικτική έναντι της Κομισιόν. Εμείς χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί στην έκθεση του εισηγητού και φυσικά προσβλέπουμε στην κατάθεση και συζήτηση των τροπολογιών και την περαιτέρω επεξεργασία από την Επιτροπή σας που πιστεύω θα είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για την περαιτέρω ανάπτυξη του για την επεξεργασία μάλλον του θέματος αυτού στην Επιτροπή Καθήλη Αρμόδια που είναι η Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπένιον για να κλείσουμε τη συζήτηση και φυσικά ο κύριος Μπένιον ε, αντικαθιστά τον εισηγητή γνωμοδότηση τον κύριο Ντεμπάκερ. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τα σχόλια των ε, σκιωδών και της ε, Επιτροπής. Από ό,τι φαίνεται ε, θα καταλήξει επικοδομητικά όλη αυτή η ιστορία. Θα ήθελα μόνο και εγώ να καταθέσω κάποιες τροπολογίες. Υπάρχουν ένα-δύο θέματα στα οποία η έκθεση αλλά και η πρόταση της Επιτροπής είναι δύσκολο να συμβιβαστούν με τους λιμένες του Ηνωμένου Βασιλείου που ανήκουν πλήρως ε, στον ιδιωτικό τομέα. Δεν ανήκουν ε, ε, στην τοπική αυτοδιοίκηση ή στις αρχές λιμένων. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο οι λιμένες βρίσκονται σε έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους. Δεν μιλάω τώρα για ε, τις εργασιακές σχέσεις. Εγώ αναφέρομαι περισσότερο σε θέματα τιμολόγησης. Εκεί λοιπόν θα καταθέσουμε κάποιες μικρές ε, τροπολογίες γιατί επιθυμούμε να υπάρξει μια διαφορετική εξέλιξη αλλά εν πάση περιπτώσει πρόκειται πραγματικά για πολύ στοχευμένες ε, τροπολογίες που θα καταθέσουμε σε πολύ συγκεκριμένους τομείς. Ευχαριστώ κύριε Μπένιον. Οι προθεσμίες για την κατάθεση τροπολογιών. Εκπνέουν στις 19 Νοεμβρίου το μεσημέρι. Προβλέπεται η εξέταση των τροπολογιών ε, στις 5 Δεκεμβρίου και οι συμβιβαστικές τροπολογίες στις 17 Δεκεμβρίου και η τελική ψηφοφορία στην Επιτροπή μας επίσης στις 17 Δεκεμβρίου. Ακολουθεί τώρα. Α, ήρθε η πρόεδρος μας. Ναι, σας δίνω το, τον προεδρικό θόκο. Ευχαριστώ πολύ. Αλλάξαμε λοιπόν Προεδρία. Και πάλι. Και ερχόμαστε στο σημείο 14. Πρόκειται για την Οδηγία 2010. 18 λέει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω αλλαγής καθεστώτος της Μαγιότ. Το κείμενο αυτό που τον έθεσαν εμένα οι συντονιστές. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα θέμα που επήγει, αφενός από την άλλη μεριά είναι και νομικό ζήτημα. Το έδαφος της Μαγιώτς άλλαξε λοιπόν καθεστώς. Κάτι το οποίο ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2014. Η Μαγιώτ γίνεται. Ε, άκρος περιφερειακή περιοχή, ενώ πριν ήταν υπερπόντιο διαμέρισμα. Η αλλαγή αυτή στο καθεστώς της Μαγιότ έχει σαν αποτέλεσμα Μαγιότ να πρέπει να εφαρμόσει διάφορα κείμενα ευρωπαϊκής νομοθεσίας δηλαδή, Άρα πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά την γονική άδεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν υπέβαλε πρόταση ώστε να αρχίσει να ισχύει το κείμενο αυτό και αυτό ε, βάσει του άρθρου 155 της συνθήκης όπου το Συμβούλιο λαμβάνει γνώση των συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων χωρίς να χρειάζεται καν διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο θεώρησε ότι η διαδικασία αυτή, όχι για τη δικιά μας την υπόθεση, αλλά για άλλες υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την αλλαγή στο καθεστώς της Μαγιότ, κινδύνευε να οδηγήσει σε μακρές συζητήσεις σύμφωνη γνώμης τελική κτλ. Και γι' αυτό προτίμησε να αλλάξει τη νομική βάση και να ακολουθήσει το άρθρο 349 και έτσι να εξετάσει το θέμα των άκρος περιφερειακών περιοχών. Το Ευρωπαϊκό βέβαια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε πρέπει ε, κατεπηγόντως να εξετάσει το θέμα. Τώρα, την πρώτη φορά που υποβλήθηκε το πακέτο αυτό αλλαγών στο καθεστώς της Μαγιότ, που είχε να κάνει με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, θεώρησε ότι η αλλαγή αυτή της νομικής βάσης από το Συμβούλιο δεν ήταν κατάλληλη και άρα μη αποδεκτή. Το παράδοξο βέβαια είναι ότι η Επιτροπή Απασχόλησης ενώ το Συμβούλιο άλλαξε την νομική βάση, ζητείτε γνωμοδότηση από την Επιτροπή Απασχόλησης. Και βασικά για να πούμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει διαβούλευση, τουλάχιστον σύμφωνα με τις νομικές μας υπηρεσίες, γιατί αυτό προβλέπει το άρθρο 155. για να τηρηθεί και η προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου του 2014. Συνεπώς, σας προτείνω ένα τροποποιημένο κείμενο εγώ, για να αποκατασταθεί η νομική βάση, έτσι όπως την προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας βέβαια συγχρόνως και μη αγνώντας το γεγονός ότι η Μαγιότ όντως από υπερπόδιο διαμέρισμα γίνεται άκρος περιφερειακή περιοχή, για την οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε τις διαρθρωτικές της δυσκολίες τόσο στο κοινωνικό τομέα όσο και στον οικονομικό. πράγμα το οποίο δικαιολογεί την καθυστέρηση εφαρμογής της νομοθεσίας. Γι' αυτό και εξετάζουμε την αλλαγή αυτή στο καθεστώς. Το Συμβούλιο είχε ζητήσει το κατεπήγον στην προηγούμενη ολομέλειά μας. Η αντιπρόεδρό μας, η Ελίζαμπετ Σρέντερ, είχε πει να αρνηθούμε το κατεπήγον. Φαντάζομαι ότι και στην επόμενη Ολομέλεια το ίδιο θα κάνει, γιατί το Συμβούλιο, για λόγους που δεν γνωρίζω, ζήτησε και πάλι το κατεπήγον. Παρόλο που το έχει απορρίψει το Κοινοβούλιο. Τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια το απέρριψε. Αλλά το αίτημα ξανάρθε. Και εμεί θέλουμε ήσυχα και ωραία, έτσι αποφασίσαμε τουλάχιστον τον Οκτώβριο, το Δεκέμβριο να καταλήξουμε έχοντας χρόνο να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Το Συμβούλιο όμως επανήλθε όπως σας είπαμε το καταπήγον. Θέλει κανείς το λόγο εδώ. Όχι. Ωραία. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας και ευχαριστώ και την Ελίζαμπετ Σρέντερ που θα πει τα ίδια στην επόμενη Ολομέλεια όπως ακριβώς είπε και στην προηγούμενη Ολομέλεια όταν θα έρθει λοιπόν και πάλι στην ημερήσια διάταξη το θέμα αυτό. Ωραία. Φόσο δεν υπάρχουν σχόλια, προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 19 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Μόνο στα αγγλικά, με ηλεκτρονική υπογραφή. Και θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή στις 26 Νοεμβρίου ώστε να τηρήσουμε τη δέσμευση που αναλάβαμε απέναντι στο Συμβούλιο που ήταν για το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια. Πάει και αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο 16. Άνταμ Κόζα. Παρουσιάστε μας τις 20 τροπολογίες στην έκθεσή σας σχετικά με την 7η και 8η έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στρατηγική έκθεση 2013 για την υλοποίηση των προγραμμάτων της περίοδου 2007-2013. Παρακαλώ κύριε Κόζα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πολύ χαίρομαι που μπορώ να μιλήσω για το κείμενο αυτό. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Έρη και τον ευχαριστώ που με αντικατέστησε μάλιστα και την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, από την τελευταία φορά μέχρι σήμερα έχουμε 20 τροπολογίες, τις οποίες κοίταξα, ανάλυσα και τις αντιμετωπίζω πραγματικά θετικά. Πιστεύω ότι όλες οι τροπολογίες ακολουθούν τον ίδιο δρόμο με μένα. Οπότε, συμφωνώ με τις τροπολογίες αυτές. Μπορώ επίσης να σας πω ήδη από τώρα πως πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και έτσι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο αυτό πολύ γρήγορα. Επιτρέψτε μου όμως παρόλα αυτά να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που μοιάζουν μεταξύ τους και οι οποίες αναφέρονται στην ίδια ομάδα ανθρώπων αλλά με διαφορετική διατύπωση για να περιγράψει ακριβώς αυτή την ομάδα ανθρώπων. Αυτό θέλω να το συζητήσω με τους σκιώδεις την επόμενη φορά, ώστε να μιλάμε την ίδια γλώσσα μεταξύ μας. Εντός εγωγικών βέβαια. Τροπολογία αριθμός 1. Μάρκιν. Θέλω να ζητήσω από την κυρία Μάρκιν να μου εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί με τη διαφορά ανάμεσα στις χώρες που αποτελούν μέρος του προγράμματος και εκείνες που δεν αποτελούν μέρος του προγράμματος. Ποια είναι αυτή η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες. Αλλιώς όλα τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνω και όλες τις άλλες τροπολογίες και όπως σας είπα μπορώ να τις δεχτώ. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή, θέλω να καταλάβω, ανάμεσα στις χώρες που αποτελούν μέρος του προγράμματος και αυτές που δεν αποτελούν μέρος του προγράμματος. Υπάρχει και μια άλλη τροπολογία της κυρίας Παπαδοπούλου, η οποία αναφέρεται σε διαφορετικές χώρες. Νομίζω ότι ίσως θα ήταν προτιμότερο να μιλάμε για περιφέρειες εδώ, για περιφέρειες ή για ζώνες του Νότου και ζώνες του Βορρά που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής. Αυτά, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ποιος θα ήθελε να λάβει το λόγο. Θέρκας και Χάρκιν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ξενομότος της κυρίας Παπαδοπούλου που δεν είναι παρούσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον κύριο Κώσα για την εργασία του και για την θετική στάση που έχει δείξει εναντί όλων των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί, των 10 τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Δεν ξέρω αν θα σταθεί η κυρία Χάρκιν, αλλά κυρίε κυρία νομίζω θα ήθελε να απαντήσει για το γεγονός ότι υπάρχουν περιοχές όπου όλες οι περιφέρειές τους καλύπτονται και εμπλέκονται σε προγράμματα αρρωγής λόγω αυτών των προγραμμάτων αρρωχής έχουμε το πρόβλημα ότι μπορούν να υπόκεινται σε κυρώσεις οι οποίες θα εμποδίσουν την παροχή διαρθωτικών πόρων. Αυτό μπορεί να αφορά ολόκληρες χώρες οι οποίες βρίσκονται σε προγράμματα αρρωγής. Γι' αυτό έχει νόημα να μιλήσουμε για περιοχές προφανώς, αλλά και για χώρες οι οποίες ως χώρες υποβάλλονται σε περιορισμούς λόγω μνημονίων σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση από τα προγράμματα συνοχής. Και τέλος, κύριε Κώσα, θα ήθελα να σας πω ότι η δική σας ε, γενεοδορία δεν πρέπει να σας επιτρέψει να δεχτείτε τροπολογίες οι οποίες είναι φανερά εκτός της ε, αρμοδιότητας της Επιτροπής μας. Οι τροπολογίες 18, 20 και 24 της κυρίας Σεσά, για παράδειγμα χάρη, ή θα πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι μη παραδεκτές γιατί είναι έξω από την αρμοδιότητα της Επιτροπής μας ή απλώς πρέπει να απορριφθούν γιατί ξεκινά μια συζήτηση για την πράσινη ενέργεια και άλλα θέματα που είναι τελείως εκτός από τις αρμοδιότητες της αρμοδιότητας επιτροπής μας. 18, 20, 24, ίσως και η γραμματεία θα πρέπει να εξετάσει αυτές τις τροπολογίες που εγώ πιστεύω ότι είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της επιτροπής μας. Συγγνώμη, η βοηθός μου λέει ότι αυτές οι τροπολογίες είναι για την επόμενη έκθεση. Συγγνώμη. Όλοι, όλοι, όλοι σφάλουμε. <clears throat> Δίνω το λόγο στην κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο Κόζα. Μου κάνατε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά στην τροπολογία υπαριθμών 1. Νομίζω ότι ο κύριος Σέρκας ε, ε, απάντησε εν μέρη Υποθέτω λοιπόν, ε, κοιτάγοντας την έκθεση από την Επιτροπή, ε, τη στρατηγική αυτή έκθεση και αναφέρεται με απόλυτη σαφήνεια ότι το σοκ της ε, κρίσης δεν έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεν το αισθάνονται έτσι οι πολίτες στα κράτη-μέλη, κυρίως σε αυτά που βρίσκονται υπό προγράμματα, έχουν πρόβλημα συγχρηματοδότησης, εξυγίανσης των χρηματοοικονομικών. Ίσως λοιπόν ίσως ε, να μην ενδείκνεται εδώ, να πρέπει κάπου αλλού. Εγώ θέλω να το συζητήσουμε, είμαι ανοιχτή. Πιστεύω όμως ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε. Και όπως είπε και ο κύριος Σέρκας, ε, υπάρχει και η απειλή των ε, κυρώσεων, παπιλούνται κυρώσει. Αυτό βέβαια είναι και αυτό άλλη ιστορία. Εγώ θέλω να αφαιρθώ στην δική μου την τροπολογία, την υπαριθμόν 16. Στη γνωμοδότησή σας αναφέρεστε σε μέρημνα για τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία. Εγώ θέλω να διαγραφεί αυτό και να αναφέρετε γενικά το θέμα της φροντίδας και των ατόμων που την παρέχουν. Ε, το ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Η κυρία Σουέτερο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Κοιτάξτε, ε, περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση, διότι βεβαίω η πολιτική συνοχή αυτή τη στιγμή δέχεται επιθέσεις. Αυτό το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε επίσης ότι ενδέχεται να υπάρξει μακροοικονομική αιρεσιμότητα για την πολιτική συνοχή. Σε αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η συνοχή και η μακροοικονομική αιρεσιμότητα ε, συγκρούνται. Η μία αποκλεί την άλλη. Εάν λοιπόν επιθυμούμε κονδύλια πράγματι να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των περιφερειών, τότε δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ε, αλληλοκατάργησης ή να χρησιμοποιούνται ως ένα είδος απειλής. Και οι εκθέσεις αυτές αποδεικνύουν πού ακριβώς υπάρχει επιτυχία, αλλά και πού ακριβώς ε, δεν υπάρχει επαρκής υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου θα εγκρίνουμε το μεγάλο πακέτο και νομίζω ότι ε, σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξετάσουμε την έκθεση, ακόμα και αν περιλαμβάνει αναδρομικά στοιχεία. Κύριος Μπουμπικό για την Κομισιόν. Ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή να σταθούμε στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι όλο το έγγραφο αυτό και η έκθεση προόδου και το στατιστικό έγγραφο έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα στην έκθεση πρόοδου αναλύουμε την κατάσταση, ενώ στο στρατηγικό έγγραφο έχουμε μια σειρά προτάσεων και συνοψίζουμε την ε, συμβολή της πολιτικής συνοχής για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει από την οικονομική κρίση. Είναι σαφές ότι καθώς βγαίνουμε από την κρίση, την ύφεση, ο αντίκτυπος της κρίσης δεν ήταν ισόμορφος σε όλα τα κράτη-μέλη, ήταν ανισομερής και φυσικά δεν έχει πάψει να υπάρχει αυτός ο αντίκτυπος. Έχει μειωθεί η σύγκληση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά το επίπεδο ανεργίας. Έχουν περιοριστεί οι δυνατότητες των κρατών μελών και των τοπικών κυβερνήσεων να προχωρούν σε συγχρηματοδότηση και να έχουν ένα λογικό επίπεδο δημοσίων επενδύσεων, κάτι το οποίο δυσκολεύει την ε, επίλυση πολλών προβλημάτων και αυτό είναι κάτι το οποίο αναφέρεται στο έγγραφο. Και φυσικά υπάρχει και ένα πρόβλημα με την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών, ιδίως στις αστικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά και αυτό προσπαθεί να προωθήσει η Κομισιόν με τις πολιτικές της, με το Ταμείο Συνοχής. Για την μακροαιρεσιμότητα που έχει αναφερθεί, η θέση της Κομισιόν είναι ότι η πολιτική συνοχή δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα σε ένα υγιές μακροοικονομικό περιβάλλον. Έχουμε λάβει υπόψη την γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά. Εξακολουθούμε όμως να έχουμε τη μακροοικονομική ελεσιμότητα στην πρότασή μας. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας σχετικά. Μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε και τη μακροαρεσιμότητα αλλά και την έννοια της αναλογικότητας στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Φέρκας Εν συντομία, πρέπει όμως να απαντήσω σε αυτά που λέει η Κομισιόν. Μου φαίνεται πάρα πολύ ανησυχητικό ότι αυτοί ακριβώς οι οποίοι θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα ενεργοί στην υπεράσπιση της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν την ε, συνοχή στην υπηρεσία της μακροαιρεσιμότητας και όχι το αντίθετο. Το να χρησιμοποιούμε λέξεις δεν επιτρέπει να χάσουμε την πραγματικότητα. Η μακροαιρεσιμότητα σημαίνει ότι οι περιοχές που έχουν υψηλή ανεργία και έλλειψη, έλλειψη ε, χρηματοδότησης θα χάσουν τη χρηματοδότηση όχι 100% αλλά 50% και αυτή είναι η γενοδορία της Επιτροπής. Ναι, κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο, ο εισηγητής. Α, συγγνώμη, κυρία Χάρκιν προηγουμένως. 30 δευτερόλεπτα, λέει η κυρία Χάρκιν. Και εγώ θέλω να υποστηρίξω απόλυτα τον κύριο Θέρκα. Σα ευχαριστώ. Κυρία Κώσα. Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Σρέντερ και με την άποψη του συναδέρφου Σέρκας. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι τροπολογίε οι περισσότερε τουλάχιστον, αντικατοπτρίζουν αυτήν ακριβώς την άποψη. Ευχαριστώ και την κυρία Χάρκιν για την απάντησή τη σχετικά με την τροπολογία αριθμό 1. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και όσον αφορά την τροπολογία 16, επαναλαμβάνω αυτό που είπα. Ότι το ίδιο πράγμα σκεφτόμαστε, για το ίδιο πράγμα μιλάμε, αλλά για μια κάπως διαφορετική πτυχή. Οπότε τελικά πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε μια συμφωνία. Περιμένω λοιπόν τώρα και προσβλέπω στη συνεργασία με τους συναδέρφους και είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε σε καλές λύσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ωραία, θα εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες στις 25 Νοεμβρίου και την επομένη στις 26 του μηνός η Ρέγγι θα αποφανθεί και 22 και μετά θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο σημείο 14. Στην έκθεση του David Κάζα, που δεν είναι όμως εδώ, τον αντικαθιστά κάποιος. Α, ο κύριος Κοζά τον αντικαθιστεί, ωραία. Πρόκειται για τις 25 τροπολογίες στην έκθεση πρωτοβουλίας του κυρίου Κάζα για ένα πλαίσιο για πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτο 2030. Είναι γνωμοδότηση τη δικιά μα Επιτροπής Στι επιτροπέ ΕΝΒΙ και ΙΤΡΕ, οι οποίες αυτές είναι αρμόδιες όσον αφορά τι δικέ τους αρμοδιότητες βάσει του άρθρου 51. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ναι, αντικαθιστώ εδώ τον κύριο Κάζα και θα προσπαθήσω να σας περάσω το δικό του μήνυμα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τους συναδέρφους για τη συνεργασία τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους σκιώδες εισηγητές και όσους υπέβαλαν τροπολογίες. Ο κύριος Κάζα πιστεύει ότι περισσότερες από τις τροπολογίες αυτές θα γίνουν αποδεκτές, μια που ακολουθεί το πνεύμα του εισηγητή. Συνεπώς, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλές συμφωνίες. Ο ίδιος έχει ήδη ετοιμάσει πέντε συμβαστικές τροπολογίες. Θα τις στείλει σήμερα το βράδυ στους σκιώδες εισηγητές ή το αργότερο αύριο το πρωί. Οι τροπολογίες 1, 2, 10, 11 και 13 και 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 είναι οι τροπολογίες οι οποίες θα καλύπτονται από τις συμβαστικές του κύριου Κάζα. Νομίζω ότι η αναλογία είναι πολύ καλή. Όσον αφορά τις τροπολογίες 3, 4 και 6, ο κύριος Κάσα μπορεί να τις δεχτεί. 5, 16, 17 και 18 για τις τροπολογίες αυτές είναι μάλλον σύμφωνος, οπότε θα συμπεριλάβει ένα τμήμα τουλάχιστον των τροπολογιών αυτών στις συμβαστικές του τροπολογίες. Συνεπώς προβλέπει ο κύριος Κάζα στη συνεργασία με τους συναδέρφους και είναι σίγουρος ότι θα μπορέσει να καταλήξει σε ένα ισορροπημένο κείμενο έτσι. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Ποιος θέλει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Σέρκας. Ναι, σύντομα και εγώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τα όσα μας είπε ο κύριος Κόσακ για τις συμβαστικές τροπολογίες που περιμένουμε σήμερα το βράδυ. Τώρα, πριν μπέρδεψα την έκθεση Κάσα με την έκθεση Κόζα. Τώρα εξετάζουμε την έκθεση Κάζα. Οπότε υπάρχουν τροπολογίες 18, 20 και 24 που δημιουργούν πρόβλημα όσον αφορά την επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Κύριε Κόσκα, σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστήστε και τον εισηγητή Κάσα εκ μέρους μας. Πρόεδρος. Ωραία. Όλα αυτά διευκρινίζονται μεταξύ Κόζα Κάζα. Εντάξει. Τώρα είμαστε εντάξει όμως, έτσι τα έχουμε ξεκαθαρίσει όλα τα ζητήματα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Ή όχι. Όχι. Τώρα ή ποτέ. Ε? Ωραία. Τώρα. Παρακαλώ. Sorry. you very much. Um, Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει στις αρχές του 2014 να έρθει με μια πιο συγκεκριμένη πρόταση όσον αφορά το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια. Το πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό. Και γιατί, γιατί συνεχίζει να στηρίζει τις πράσινες τεχνολογίες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Προς το παρόν ετοιμάζουμε μια έκθεση αξιολόγησης όπου επιπτώσεις επί της απασχόλησης λαμβάνονται πλήρως υπόψη. Όσον αφορά τα 5 εκατομμύρια στοιχεία από πλευρά Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας. Ξανακοιτάμε όμως τι επιπτώσεις μακροπρόθεσμα των πολιτικών κλίματος και ενέργειας πάνω στην απασχόληση. Τι θα βγει από τη συνεχιζόμενη έκθεση αξιολόγηση είναι, πιστεύω, μία αλλαγή σε τομείς που επηρεάζουν την απασχόληση και στην κατάρτιση και η απασχολησιμότητα πρέπει πλήρως να ληφθεί υπόψη. Ε, σας ευχαριστώ ε, κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πρέπει να είσαστε απόλυτα γαλήνια γιατί θα δώσω όλα τα μηνύματά σας στον κύριο Κάσα και χαίρομαι που μπορώ να δω ότι όλες οι τροπολογίες είναι στη σωστή θέση. Μπορούμε να κλείσουμε με το σημείο αυτό της ημερησίας. Εντάξει, οι βασικές τροπολογίες θα εξεταστούν στις 17 Δεκεμβρίου και θα ψηφιστούν ως Νούπο την ίδια μέρα, ώστε να μπορέσουμε να γνωμοδοτήσουμε εγκαίρως στις Επιτροπές Ήτρα και ΕΝΒΙ που θα ψηφίσουν στις 9 Ιανουαρίου πριν από την Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Το τελευταίο σημείο της σημείωσης διάταξης είναι τα πεπραγμένα της Επιτροπής της Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων που πήγε στην Κροατία στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Μία αντιπροσωπεία στην οποία δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω αλλά τις οποίες ηγήθηκε ο κύριος Τσάβα Όρη και που τον βοήθησε η Έντιτ Bauer για τη σύνταξη των πεπραγμένων. Κύριε Μπάουερ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Προσπαθώ και εγώ να μιλήσω εν συντομία. Εγώ δεν ήμουν το πιο σημαντικό μέλος αυτής της αντιπροσωπείας. Ο κύριος Έρη ήταν αυτός, ο οποίος ήταν βέβαια και είχε τον κύριο Φίλιπ Μπουλάν μαζί του και την Ρουζάν Τόμασίτς από το ECR. Μια μικρή ομάδα λοιπόν βουλευτών πήγε στην Κροατία, στο Ζάγκρεπ, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2013. Δύο σημαντικές παρατηρήσεις μονάχα έχω να κάνω. Καταρχήν ότι μεταξύ των νέων η ανεργία φτάνει το 50% είναι το τρίτο χειρότερο αποτέλεσμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης άμα κοιτάξουμε την κατάσταση των νέων στην Κροατία, τα 80% των νέων δεν έχουν πραγματική εργασία, έχουν μονάχα περιστασιακές θέσεις εργασίας, έχουν <clears throat> συμβάσεις περιορισμένου χρόνου. Η Κροατία λοιπόν Προσδοκάμε με την πρωτοβουλία για τους νέους. Όλα αυτά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους νέους, μεταξύ των οποίων και η εγγύηση για τους νέους θα είναι πολύ σημαντικά για την Κροατία. Αυτή είναι η πρώτη μας διαπίστωση. Η δεύτερη είναι ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντική η μαύρη εργασία. Ενεκρίτη πρόσφατα νομοθεσία σε σχέση με τους εποχιακούς εργαζόμενους. Η κατάσταση των εποχιακών εργαζομένων στη Γεωργία έχει καλυφθεί σε νομικό επίπεδο, έχουν νομιμοποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ υψηλή υψηλό το ποσοστό μαύρης εργασίας που είναι περίπου 30%. Μιλήσαμε με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και μας είπαν ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό αυτό σε ορισμένου τομεί όπου μπορεί να φτάσει το 60% η μαύρη εργασία. Ιδίω στην παροχή υπηρεσιών. Η Κροατία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να προχωρήσει σε μια μεταρρύθμιση του εργασιακού της δικαίου και φυσικά θα πρέπει να εργαστεί και να αγωνιστεί κατά της ε, μαύρης και φαιάς εργασίας. Μια τελευταία παρατήρηση. Ήταν κάπως παράδοξη η μορφή της επισκεψής μας, γιατί η Κροατία βρισκόταν τότε σε διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ορισμένα άλλα θέματα και δεν υπήρξε ιδιαίτερη ικανοποίηση να, σε ό,τι αφορά την υποδοχή της ε, μας. Υπήρξε μια διαμάχη με κάποιον ε, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Κροατίας, ο οποίος κατηγορείται για πολύ σοβαρά δικήματα και δύο μέρες μονάχα μετά πριν από την ένταξη της ε, Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελήφθη μια απόφαση για τη χρήση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης όπου η Κροατία απέρριψε την χρήση αυτού του εντάλματος. Όλα αυτά είχαν μεγάλη απήχηση στα μέσα ενημέρωσης στην Κροατία. Λόγω όλων αυτών των γεγονότων το κλίμα δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικό σε ό,τι αφορά την αντιπροσωπεία μας στην Κροατία. Επίσης, Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την κατάρτιση των νέων στην πληροφορική. Πρόκειται για ένα μικρό μονάχα αριθμό ατόμων, καμιά σαρανταριά άτομα, αλλά είναι ένα σημαντικό εγχείρημα το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία μεταξύ των νέων και απλώς σας το λέω αυτό για να μπορέσω να πω κάτι το θετικό, ότι πράγματι υπήρχαν και ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να λάβει το λόγο. Όχι, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Edith Bauer για την ε, ε, έκθεση πεπραγμένων στην Κροατία. Νομίζω λοιπόν ότι έχει τελειώσει η μέση διαταξή μας γιατί κανείς δεν θέλει να λάβει το λόγο σε σχέση με τα διάφορα σημείο 19 και θα τα ξαναπούμε στις 18 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο θα είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η ψηφοφορία που θα κάνουμε στις 7 η ώρα, στις 18 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο και μετά στις 21 Νοεμβρίου. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε μια κοινή συνάντηση την 5η ε, το πρωί με την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή για να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση από τον κύριο Όλη Ρεν, εκ μέρους της Επιτροπής της έκθεσης για την ε, ανάπτυξη και του μηχανισμού Έγκυρης προειδοποίησης που δημοσιεύτηκε χθε από την Κομισιόν και άλλες δύο συνεδριάσεις θα κάνουμε στις 25 και 26 Νοεμβρίου και το απόγευμα της πρώτης και το πρωί της Δευτέρας αλλά έχω προχωρήσει με μεγάλη ταχύτητα, υπερβολική ταχύτητα και η κυρία Ρέιντερς θέλει να θέσει ένα θέμα χαρακτήρα διαφόρου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο αγαπητοί συναδέλφου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να γράψω για τα πρακτικά ε, ότι λυπάμαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι η Επιτροπή αυτή συνεδριάζει ειδικά κατά τη διάρκεια της ε, εβδομάδας ε, των πολιτικών ομάδων. Ε, ξέρω ότι υπάρχουν βέβαια λόγια ότι το κάνει αυτό, αλλά μην ξεχνάτε και το επισημένο για άλλη μια φορά. Αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη ειδικά στις πολιτικές ομάδες. Παρακαλώ να καταγραφεί. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταλαβαίνω απόλυτα τις ανησυχίες σας. Αν πάρετε όμως τον πίνακα αυτών που έχει χαρακτήρα αναδέλτου κοινοβουλευτικών εργασιών αναφέρεται ότι η σημερινή μέρα είναι μια μέρα η οποία είναι διαμεμοιρασμένη μεταξύ κοινοβουλευτικών εργασιών και εργασιών των πολιτικών ομάδων. Αυτό δεν ε, γίνεται για άλλο λόγο παρά για να εξασφαλίσει ότι οι βουλευτές μπορούν να βρεθούν και εκτός της έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν αυτούς οι οποίοι παρακολούσαν τη σημερινή συνεδρίαση, ιδίως αυτούς που έμειναν μέχρι το τέλος. Και όταν εγκρίνουμε την ε, ημερήσια διαταξή μας για το 2014 μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν τέτοιες ε, ε, περιπτώσεις, αλλά αυτό έχει να κάνει με την μορφή της οργάνωσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επομένως η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές ομάδες και τις επιτροπές επέλεξε να υπάρχει αυτή η επικάλυψη επιτροπών και πολιτικών ομάδων. Δεν φταίω εγώ λοιπόν. Σας ευχαριστώ και σας δίνω ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα το βράδυ στο Στρασβούργο, σε 7 η ώρα.